Se prendete posto possiamo cominciare i nostri lavori. Εάν καθίσετε μπορούμε να ξεκινήσουμε. pomeriggio riprendiamo con... Eh, Τώρα το απόγευμα θα συνεχίσουμε την ακρόαση για το πακέτο που αφορά τα ταξίδια. Οδηγία πάρα πολύ σημαντική διότι αφορά κυρίως ε, εκατομμύρια χρήστες που είναι και οι καταναλωτές το σημείο αναφοράς αυτής της ε, οδηγίας, της ε, Επιτροπής, συγγνώμη. Για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, χρόνο που χάνουμε συνήθως σε τέτοιου είδους περιστάσεις, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, εισηγητή μιας έκθεσης, την οποία θα συζητήσουμε κάποια στιγμή ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο στον Hans Peter Mayer. Μετά από τον κύριο Μάγερ, τον λόγο θα πάρει εκ μέρους της Επιτροπής ε, Μεταφορών που γνωμοδοτεί για αυτή την οδηγία ο κύριος Ισμαήλ Έρτοκ, τον χαιρετώ και αυτόν. Και ξεκινάμε με τον Χάνς. Χάνς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Έχουμε σημαντικό θέμα ενώπιον μας και έχει γεννήσει και μεγάλο ενδιαφέρον. Αντίστοιχα με τα δικαιώματα των επιβατών που εγκρίναμε το πρωί και να σας πω τι έγινε εκεί. Ψήφισε πρώτα η δική μας επιτροπή, γιατί επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Μεταφορών και στην τωρινή οδηγία την παρούσα που μας απασχολεί τώρα, που είναι τα οργανωμένα ταξίδια, είναι ακριβώς το αντίθετο. Γνωμοδοτεί η Επιτροπή Μεταφορών και εμείς έχουμε τον τελευταίο λόγο γιατί είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας. Και μηδιώντας λέω ότι όλα εδώ πληρώνονται, ότι πραγματικά τα του Κέσσαρου στον Κέσσαρη, το αλλά αυτό το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι τα δικαιώματα των επιβατών. Γιατί με τους επιβάτες έχουμε μια πτήση από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, αν θέλετε και με τα αποκρίσεις. και τελειώνει η υπόθεση. Εδώ έχουμε πολλούς ε, ενεχομένους που παρέχουν υπηρεσίες, ε, που προσφέρουν διάφορα ε, και μπορούν να συμβούν επίσης διάφορα. Και ο στόχο δεν είναι μεταφορά από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, αλλά ο σκοπό είναι να περάσει κανεί ευχάριστε διακοπέ. Και όταν υπάρχουν κάποια επεισόδια και περιστατικά αξιολογούνται πολύ διαφορετικά, ε, όπως και οι επιπτώσεις τους, από ότι σε μια απλή πτήση. Είναι λοιπόν μεγάλο το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και αυτό φαίνεται και από τις θέσεις και τα έγγραφα θέσεων που μας έχουν στείλει. Πάρα πολλά email λαμβάνουμε και πολλοί ζητούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Ε, θα προσπαθήσω να τα αποκριθώ σε όλους, να έχω και επαφέ και συνομιλίες με τους ενεχομένους. Για μας αυτό είναι προφανές και αυτονόητο άλλωστε. Σε αντίθεση ε, με κάποια εθνικά ήθη ε, που θεωρούν αρνητικό το λόμπι, εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ε, οπωσδήποτε και πάρα πολύ να μας πιέζουν οι ενδιαφερόμενοι γιατί όταν νομοθετούμε και αφορά τη ζωή τους αυτό πρώτο μας καθήκον είναι να ακούμε αυτούς που θίγονται από την νομοθεσία για να δούμε τι είναι εφικτό, ε, τι δεν είναι και να μην τους παραγωνίζουμε και να τους χαρακτηρίζουμε ομάδες πίεσης. Υπάρχει μια πρόταση ε, και νομοθεσία ε, της δεκαετίας του 90 και θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Στο μεταξύ έχουν ε, αλλάξει πολλά, αρκεί να αναφέρω και μόνο το διαδίκτυο. Επίσης χρειάζεται κάποια προσέγγιση και ε, με την οδηγία για τα δικαιώματα των επιβατών που ψηφίζαμε σήμερα το πρωί και προσεχώς η Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει όλες αυτές οι ρυθμίσεις να είναι κατανοητές, εύληπτες και φιλικές προς το χρήστη. Αν δείτε τη σημερινή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θα καταλάβετε ότι πολλές προτάσεις πρέπει να τις διαβάζετε ξανά και ξανά, πολλές φορές μέχρι να καταλάβετε τι θέλει να πει ο ποιητής. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας. Και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ένα ισόρροπο αποτέλεσμα ε, και να συγκεραστούν και τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα των ε, επιχειρήσεων και των ε, πελατών. Δεν πρέπει να μείνουν δυσαρεστημένοι ή ικανοποιημένοι οι δε. Θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο για να μπορούν να συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις και να πηγαίνει ο κόσμος διακοπές. Ε, η ανωτέρα βία, η προστασία από την αφαιρεκιότητα, η αστική ευθύνη, οι ε, αυξήσει των τιμών, οι προθεσμίες, όλα αυτά και άλλα πολλά ακόμα είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν. Ε, και με χαρά θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας και χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει με ερωτήσεις και απαντήσεις. Και σας παρακαλώ να κάνετε και ερωτήσεις όλοι και όχι απλές δηλώσεις για να μην ανατραπεί το χρονοδιάγραμμα και ε, το πρόγραμμα. Λοιπόν, πρώτα παρουσιάσεις, μετά έρωτα αποκρίσεις. Ε, σταματώ εδώ και ξαναδίνω το λόγο στον Πρόεδρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Μάγερ και δίνω το λόγο για τη, στην Επιτροπή Μεταφορών και στον κύριο Χέτζοκ. Yes, thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Στα αγγλικά. Ζητεί συγγνώμη ο συνάδελφος Λιπεράτσκι, ο οποίος είναι εισηγητής, είναι εισηγητής αυτού του σημαντικού θέματος και δυστυχώς σήμερα κολλείται και δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική ακρόαση. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι είναι σημαντικό το θέμα και μας ενδιαφέρει πολύ ως Επιτροπή Μεταφορών, ακριβώς γιατί έχουμε ε, όλες αυτές τις αρμοδιότητες για τις μεταφορές, του τουρισμό και τα δικαιώματα ε, των επιβατών. Να σας πω λοιπόν τι λέει ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ε, οι καταναλωτές χρειάζονται προστασία ιδιαίτερη όταν ταξιδεύουν. Γι' αυτό εγκρίθηκε και η αντίστοιχη οδικία το 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια. Έκτοτε έχει αλλάξει πολύ ε, με το επιγραμμικό εμπόριο η κατάσταση αλλά και με την απελευθέρωση των αερομεταφορών. Και ο κόσμος ε, οργανώνει τις διακοπές του με διαφορετικό τρόπο από τη δεκαετία του 90. Όλο και περισσότερο οι καταναλωτές είναι πιο δραστήριοι ε, στο να σχεδιάζουν τις διακοπές τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με το διαδίκτυο. Δεν επιλέγουν δηλαδή από πακέτα που είναι ήδη έτοιμα, αλλά το ε, κόβουν και το ράβουν στα μέτρα τους το κάθε πακέτο. Αυτό οδηγεί σε αυξανόμενη ανασφάλεια για το ποια ε, κατάσταση επικρατεί και πώς θα μπορούν να επωφελούνται ε, οι καταναλωτές και τι ισχύει για αυτούς. Πολύ συχνά οι καταναλωτές αγνοούν καν τη δυνατότητα προστασίας που έχουν και τι μπορούν να αναμένουν σε κάθε δεδομένη κατάσταση. Θα πρέπει βεβαίως η νομοθεσία να ενημερωθεί για να καλύψει κάποια σχήματα πωλήσεων που δεν υπήρχαν όταν εγκρίθηκε το 1990. Ο συνεισηγητής έχει τους εξή στόχους. Πρώτον, η νέα οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίζει ε, όφελος των καταναλωτών και να ε, έχουν υψηλή προστασία όταν συνδυάζουν ένα πακέτο ε, υπηρεσιών. Ε, στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού για όλους ε, χωρίς ε, νομικά εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόδιο ε, και να τα τηρούν όλα αυτά επιχειρήσεις ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής. Οι ορισμοί τις οδηγίες θα πρέπει να διευκρινιστούν γιατί η αγορά εξελίσσεται πιο γρήγορα από την νομοθεσία και θα πρέπει οπωσδήποτε να ορίσουμε ποιος συνδυασμός επιγραμμικών ή μη υπηρεσιών θα καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογή της παρούς οδηγία. Μπορεί κανείς να πει ότι το πεδίο εφαρμογή της οδηγία δεν είναι αρκετά ευρύ, γιατί τα οργανωμένα πακέτα είναι όλο και πιο ξεπερασμένα. Από τότε που εγκρίθηκε το 90 λοιπόν αυτή η αγορά έχει αλλάξει πολύ και η προτίμηση και η συμπεριφορά των καταναλωτών ε, με τρόπο ραγδαίο. Ας πούμε, οι μεμονωμένες συμβάσεις εξαιρούνται ρητά από την οδηγία και μόνο οι συνδυασμοί υπηρεσιών όπως είναι πακέτα και ATA που είναι κάποιες ρυθμίσεις με παροχή συνδρομής στον τόπο των διακοπών. Ε, ελάχιστες λοιπόν προδιαγραφές για εναρμόνιση αλλά και πάλι η οδηγία δεν δίνει σαφή καθοδήγηση για το αν είναι κατελάχιστο ή καταμέγιστο αυτή η μεγιστο αυτη η εναρμονιση Σε ποιο βαθμό λοιπόν θα εναρμονιστεί αυτό και γιατί επέρχεται ε, νομική ανασφάλεια. Η πλήρη εναρμόνιση σημαίνει ενιαία και ομοιόμορφη προστασία των καταναλωτών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμποδίζει τα κράτη-μέλη όπου χρειάζεται να ε, εγκρίνουν πιο ευνοϊκά μέτρα για τους καταναλωτές, όπως συμβαίνει με τη σημερινή οδηγία για τα οργανωμένα ε, ταξίδια. Αυτή είναι μια πολιτική και μια επιλογή που θα πρέπει να ε, αποφασιστεί από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Όποια πάντως απόφαση να ληφθεί, το επίπεδο εναρμόνισης θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο της οδηγίας, σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη η πρόταση ορίζει ότι ο διοργανωτής και όχι ο λιανέμπορος του πακέτου ε, θα πρέπει να φέρει την αστική ευθύνη, ο tour operator δηλαδή, απέναντι στον καταναλωτή. Ε, ε, η νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών αφορά μόνο στο διοργανωτή και όχι τον πράκτορα που πολύ στη λιανική που θεωρείται απλώς μεσάζων ενδιάμεσος του tour operator. Παρ' όλα αυτά, η αγορά έχει συγκλίνει και σήμερα πολλές φορές ε, και τα ίδια τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες, είναι ε, οργανωτές γιατί εκείνοι φτιάχνουν τα πακέτα ε, σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή, του πελάτη. Και επίσης πολύ συχνά οι tour operators πολλούν τα πακέτα άμεσα στον καταναλωτή χωρίς να περνούν μέσα από τους παραδοσιακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Επίσης υπάρχουν και ε, περιπτώσεις ε, όπου ο tour operator ή το πρακτορείο φέρει την ευθύνη, αλλά ο καταναλωτής, ο πελάτης, ο τελικός δεν ξέρει ποιος έχει την ευθύνη και ποιον θα αποταθούν όταν υπάρχει μια διένεξη. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη του καταναλωτή να επιλύει αποτελεσματικά τα προβλήματα που μπορεί να ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των διακοπέων του. Χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο ε, συνυπευθυνότητα και του πράκτορα και του tour Η νέα βελτιωμένη οδηγία λοιπόν, δεδομένη και του, της κατακαιρματισμένης νομοθεσίας, καθώς επίσης και των ε, ραγδαίων εξελίξεων που πάντα είναι μπροστά από τον νόμο, δηλαδή πιο γρήγορα τρέχουν οι εξελίξεις από την νομοθεσία, θα πρέπει να έχουν συνολικά ε, μέτρα αντιμετώπισης οι καταναλωτές όλο και περισσότερο κινούν από την ιδέα ε, του οργανωμένου πακέτου και επιλέγουν, φτιάχνουν μόνοι τους το πακέτο ε, με επιτόπου ε, συνδρομή και παροχή κάποιων υπηρεσιών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τα νέα δεδομένα και οι περισσότερες οδηγίες προστασίας των καταναλωτών ρητά εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογή τους τον κλάδο των μεταφορών. Αυτά είναι λοιπόν τα σημεία που ήθελα να τονίσει ο συνάδελφος και εισηγητής κύριος Λιμπεράτσκι και ελπίζω να συμφωνείτε με όσα ακούσατε προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ Ισμαήλ και ευχαριστώ και τον συνάδελφο Λιμπεράτσκι που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Περνάμε στη συζήτηση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, καλεσμένους μας, ε, δηλαδή στους εμπειρογνώμονες που, που θέλησαν να συζητήσουν ε, σήμερα το απόγευμα μαζί μας. Η πρώτη καλεσμένη μας είναι η κυρία Μονή Γκογιάνς, που είναι Γενική Διευθύντρια της ΒΕΙΚ. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους ομιλητές να σεβαστούν το χρόνο ομιλίας των 10 λεπτών. Έχετε το λόγο. Μονίκη. Ευχαριστώ. Απόγευμα, ήθελα, ε, καλό απόγευμα. Θα ήθελα να κάνω μία παρουσίαση PowerPoint και ελπίζω να, την, ε, ε, να έχει φορτιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε την, ε, τους καταναλωτές. Ε, θα είμαι η φωνή των καταναλωτών στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ τα 10 λεπτά, έστω και αν δεν είναι αρκετά για να ε, παρουσιάσω όλα τα, τα σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας που αφορούν τους καταναλωτές. Τέλος πάντων, ε, η θέση μας ούτως ή άλλως έχει οριστικοποιηθεί και θα αποσταλεί τις επόμενες μέρες στα μέλη της Επιτροπής αυτής, αλλά και των άλλων ε, ενδιαφερομένων επιτροπών. Κάποια μηνύματα. Αυτή η πρόταση είναι, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο κομμάτι νομοθεσίας, όχι μόνο για το περιεχόμενό της, διότι ούτως ή άλλως υπάρχουν κάποιες ε, διατάξεις που προφανώς θα, θα βελτιώνονταν αν ήταν πιο Ε, αλλά πρέπει να συνδυαστούν και με άλλες ε, κοινοτικές νομοθεσίες, ε, το εθνικό αστικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, ε, την προστασία καταναλωτών στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων όλα αυτά τα θέματα είναι δύσκολα, δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Ξέρω ότι υπάρχει μία τάση να προωθήσουμε την πρόταση αυτή ε, μέχρι το τέλος της θητείας, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι είναι ε, καλύτερο να μην βιαστούμε, να είναι καλή η νομοθεσία παρά να ε, υιοθετηθεί γρήγορα. Διότι οι καταναλωτές θέλουν ένα σαφές και ξεκάθαρο περιβάλλον. Θα ήθελα καταρχάς να σχολιάσω αυτά τα στοιχεία που βλέπετε και στη διαφάνεια και προφανώς ε, χρειάζεται να αναθεωρηθεί η οδηγία. Ε, ε, ήδη έχουμε καθυστερήσει το πακέτο για, το, τα, για ταξίδια της δεκαετίας του 90 ήταν πάρα πολύ καλή η νομοθεσία τότε, φιλική προς τον καταναλωτή, όμως τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι προσδοκίες των καταναλωτών έχουν αλλάξει, ο τρόπος ταξιδίου έχει αλλάξει, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Γι' αυτό είναι, για τους καταναλωτές είναι κάπως συγκεχημένη η κατάσταση, διότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δεν είναι ακόμα σαφείς, κυρίως ε, σχετικά με το, λαμβάνοντας υπόψη το συνδυασμό των μέσων ε, μεταφοράς κτλ. που χρησιμοποιούν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, το πακέτο, το κλασικό πακέτο ε, ταξιδιού δεν είναι πλέον ε, αυτό το οποίο προωθείται. Έχουν, έχει γίνει μία μια έρευνα στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία κτλ και είδαμε ότι 4 στους δέκα ε, τουρίστες αγοράζουν το κλασικό πακέτο. Άρα δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις. Τώρα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η νέα πρόταση ε, λαμβάνει ή προτείνει μάλλον μια διευρυμένη ε, αντιμετώπιση των πακέτων. Όχι μόνο το κλασικό πακέτο, αλλά το ε, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του επιβάτη κτλ. Αυτό τι σημαίνει θεωρητικά ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα καλύπτονται, θα προστατεύονται από τις διατάξεις οδηγίες. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι η πρόταση προβλέπει δύο κατηγορίες συνδυασμών ταξιδιού. Το πακέτο και η υποβεηθούμενη ταξιδιωτική ε, ρύθμιση αυτή η διαφοροποίηση έχει συνέπειες, διότι για το Assisted Travel Arrangement ο πολιτής δεν έχει καμία υποχρέωση εκτός ε, για την προστασία σε περίπτωση χρεοκοπίας. Και ποιο είναι το πιο προβληματικό, ότι το, κατά πόσον, το, για το ερώτημα το κατά πόσον ε, εγώ σαν καταναλωτής ε, εντάσσομαι είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, είναι τελείως ασαφέ. Δεν ξέρει ο καταναλωτή. Και προφανώς είναι πάρα πολύ εύκολο για τους ε, πολιτές, αν θέλετε, να κάνουν μια διαφορετική παρουσίαση για να ξεφύγουν, για να ε, μην δεσμευτούν από τις ε, συγκεκριμένε και αυστηρές διατάξεις που προβλέπει το πακέτο. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα της πρότασης διότι δεν υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς το καταναλωτή. Να ξέρει αυτός ο άνθρωπος, είναι σε πακέτο ή είναι σε μια ε, κατάσταση υποβοηθούμενης, αν θέλετε, ρύθμισης ε, του ταξιδιού του. Τώρα, η προστασία σε περίπτωση χρεοκοπίας. Ε, όντως, ε, θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι προστατεύεται ο καταναλωτής από την χρεοκοπία, διευρύνεται ε, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και διευρύνεται και η έννοια του πακέτου. Ακόμα και αυτοί δηλαδή που ε, απλώς υποβοηθούνται στο ταξίδι τους, καλύπτονται από την προστασία σε περίπτωση χειροκοπίας. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα στην ε, οδηγία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν ανήκουν στο πακέτο, δεν ξέρουν ακριβώς από τι τους προστατεύει, από τι προστατεύονται, από την χρεοκοπία του πολιτή του πρακτορείου δηλαδή ή από την χρεοκοπία και των άλλων ε, ε, επιχειρήσεων με τις οποίες έχετε σε επαφή. Εδώ ε, επομένως πρέπει να υπάρξει μια νομική σαφήνεια. Όσον αφορά την ευθύνη για κακή επίδοση. Αφορά, τον, αφορά το πακέτο και είναι ο οργανωτής ο οποίος είναι υπεύθυνο. Αυτό το είπε και ο εισηγητής στην Επιτροπή ε, μεταφορών αυτό δεν ε, βοηθάει τους καταναλωτές. Ο καταναλωτής, την αυτό, το πρώτο άτομο το με το οποίο έρχεται σε επαφή είναι ο πολιτής. Αυτός έχει ευθύνη και ο πολιτής έχει και τις επαφές. Ο οργανωτής μπορεί να είναι σε μια άλλη χώρα, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχόμενα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κοινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή, δηλαδή κοινή ευθύνη οργανωτή και πολιτή. Και μετά θα πρέπει να ε, υπάρχει και μια ρήτρα διασφάλισης ανάμεσα στους ίδιους τους, ε, ε, επαγγελματίες έτσι ώστε αυτός ο οποίος είναι ουσιαστικά υπεύθυνο να αναλάβει και την ευθύνη. Ήδη υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα προστασίας ανάμεσα σε 10-13 κράτη-μέλη που λειτουργεί δηλαδή κανονικά και θα είναι μια μείωση, αν θέλετε, της προστασίας εάν η παρούσα πρόταση γίνει δεκτή. Τώρα, σε επίπεδο εναρμόνισης, είναι, πρέπει να δούμε ε, αν είναι σαφές ε, εάν προτείνεται πλήρης εναρμόνιση ή όχι. Αν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, τότε μειώνονται τα, τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών σε πολλές χώρες. Διότι υπάρχουν σε κάποιες χώρες ε, οι ελάχιστες ε, ε, ρήτρες προστασίας που έχουν υιοθετηθεί. Όμως, σε όλα τα κράτη-μέλη θα υπάρξει μία μείωση του επίπεδου προστασίας και μείωση των δικαιωμάτων. Διότι Υπάρχει παραδείγματο χάρη η αρχή ότι ο καταναλωτής ε, θα συμφωνήσει σιωπηρά σε περίπτωση ε, αλλαγή του συμβολέου. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση σύμφωνα με την πρόταση εάν ο καταναλωτής δεν αναφέρει επιτόπου, επιτόπου εκεί που βρίσκεται ας πούμε στο ταξίδι του το πρόβλημα ή, ή περιορίζεται η, η περιοριζεται η αποζημίωσής του για, σε τρεις νύχτες και 100 ευρώ ανανύχτα. νύχτα. Επομένως, εάν θελήσουμε να, να επιτύχουμε μια πλήρη εναρμόνιση, θα υπάρξει μια υπαναχώρηση στα δικαιώματα των καταναλωτών. Επομένως, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε σαφή κριτήρια, θα πρέπει οι υπάροχοι των υπηρεσιών να μην μπορούν να ξεφύγουν ε, από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους καταναλωτές. Επίσης πιστεύουμε ότι οι πολιτές των συνδυασμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει εκτός από την ε, προστασία που προσφέρουν απέναντι στη χρεοκοπία, να έχουν και άλλες υποχρεώσεις ε, ε, για, το, για τα διαβατήρια, για τα, για τα φάρμακα, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις, να διορθώσουν κρατήσεις κτλ. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει μια κοινή ευθύνη για τα, για τις, ε, για τα πακέτα, κοινή ευθύνη του πολιτή και του ε, οργανωτή. Θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να εξετάσει πολύ προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι πρόταση αυτή, διότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι δίκαιοι και οι κανόνες και οι διατάξεις των συμβολών αλλά και τις δυνατότητες υπαναχώρησης σε περίπτωση ε, πωλήσεων εξ αποστάσεων. Ε, Εμείς επίσης πιστεύουμε ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να είναι μια οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης, ε, όχι πλήρους εναρμόνισης, διότι αλλιώς θα θυγούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μίσελ Ντεμπλούστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσο φορτώνει η παρουσίασή μου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να βρίσκομαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας. Χάρηκα ιδιαίτερα όταν άκουσα το δόκτορα Hans Peter Mayer όταν είπε στη, στα εισαγωγικά του σχόλια ότι η οδηγία πρέπει να διατηρήσει μια καλή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και του καταναλωτή. Και με πολύ χαρά το λέω αυτό, γιατί είναι και ένας από τους στόχους ε, που προσπαθεί να επιτύχει ο οργανισμός μας. Να σας πω και ποιοι είμαστε. Εκπροσωπούμε στις Βρυξέλλες ε, μέσω 31 ε, οργανώσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΕΟΧ, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τους πράκτορες στο διαδίκτυο, του operators, επιχειρήσεις διαχείρισης ταξιδίων. Είναι ένας περίπλοκος τομέας, πάνω από 70.000 επιχειρήσεις επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες, 500.000 ε, ε, πολίτες ε, στις 28 χώρες μέλη εργάζονται στον τομέα αυτό. Το 2012 είχαμε τζίρο το, το 2012 192 δισεκατομμύρια από τα οποία τα 15 ήταν υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η νομοθεσία αυτή για μας ε, θα είναι η ραχοκοκαλιά ε, της ε, δουλειάς μας και η αναθεώρηση, η επιτυχής αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας θα έπρεπε να καλύπτει τρεις βασικές αρχές και χάρηκα όλος ιδιαίτερος που αναφέρθηκαν ήδη Πρώτα απ' όλα μια ισότιμη μεταχείριση μεταξύ όλων των ε, συμμετεχόντων στην αγορά, γιατί προφανώς ε, δεν υπάρχουν μόνο οι tour operators και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, αλλά υπάρχουν και πράκτορες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, ε, που πολλούν συνδυασμένες υπηρεσίες και θα πρέπει η μεταχείρισή τους να είναι ισότιμη. Δεύτερον, και συμφωνούμε με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, και η το είπε άλλωστε. Χρειαζόμαστε ένα καλό επίπεδο προστασίας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα στις διασυνοριακές πωλήσει. Τρίτον, και εξίσου σημαντικό, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ευρώπη ως προορισμός είναι σε ανταγωνισμό με, τους υπόλοιπους, με, την με τον υπόλοιπο κόσμο και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού κλάδου διατηρείται. Βλέπετε τι έχει συμβεί στον αεροπορικό τομέα με ε, την νομοθεσία εμπορίας ε, ε, εκπομπών αερίων. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά πάση περιπτώσει οι ανταγωνιστές μας τρίτων χωρών μας πίεσαν πάρα πολύ. Πού βρισκόμαστε σήμερα κυρίες και κύριοι και πού ήμασταν στο παρελθόν. Λοιπόν, όπως υπόθηκε και προηγουμένως από τον δόκτορα Μάιερ, σε 25 χρόνια ο κλάδος μετακινήθηκε από τα χάρτινα φυλάδια ε, στις ε, κινητές εφαρμογές σε λιγότερο από μία γενεά. Έχουμε λοιπόν μία... Υπάρχουν λοιπόν πολλαπλοί τρόποι ενημέρωσης και πολλαπλή τρόπη πώληση αυτών. Αυτό δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο για μας, να μπορέσουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίπλοκη κατάσταση στην αγορά. Υπό το φως λοιπόν αυτής της δύσκολης και περίπλοκης κατάστασης αγοράς θα θέλαμε να υποβάλουμε κάποιες συστάσεις στην Επιτροπή σας και ε, στους αξιότιμους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με τους ορισμούς που αναφέρονται στην οδηγία. βασικός ορισμός είναι βέβαια του ε, πακέτου, ε, του οργανωμένου ταξιδιού. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να καλύπτονται μόνο τα παραδοσιακά πακέτα που αναφέρονται για παράδειγμα σε ένα φυλάδιο, αλλά και δυναμικά ε, πακέτα. Ε, μπορεί δηλαδή ο καταναλωτής να πάει στο διαδίκτυο και να μπορέσει να ε, φτιάξει ένα ταξίδι με συγκεκριμένα αεροπορικά ταξίδια και διαμονή και επίση συναλλαγές που θα είναι βέβαια πολύ πιο εύκολες για τον καταναλωτή όταν ε, από έναν ιστότοπο αγοράζει μια υπηρεσία και μετά πηγαίνει μέσω αυτού του ιστοτόπου σε έναν άλλο ιστότοπο από τον οποίο αγοράζει κάτι άλλο. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι τμήμα του ορισμού του πακέτου. Αυτό το οποίο συμβουλεύσαμε τον νομοθέτη να κάνει είναι να ε, εξαιρέσει τις ε, τα ταξίδια για ε, επαγγελματικούς λόγους, γιατί αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας, ε, οπότε το νομικό πλαίσιο ε, εντός του οποίου λαμβάνει η χώρα είναι εντελώς διαφορετικό. Παρατήρησα, παρακολούθησα με ενδιαφέρον τα σχόλια του κυρίου Χέρτουκ σε σχέση με το επίπεδο εναρμόνισης και θα θέλαμε να κάνουμε μία σύσταση, κύριε Πρόεδρε. Θα προτείναμε λοιπόν στον νομοθέτη να δει τι στόχο, ε, τι, τι εννοούμε ε, εναρμόνιση, ποιος είναι ο στόχος μας. Υπάρχει νομοθεσία που δεν είναι εναρμονισμένη σήμερα. Ε, η οδηγία του 90 έδωσε δυνατότητα σε διαφορετική εφαρμογή από τα διάφορα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε όμως πλέον η εφαρμογή να είναι πιο αποτελεσματική σε επίπεδο κράτους-μέλους, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ε, περισσότερη ευελιξία στην εφαρμογή όσον αφορά, για παράδειγμα, την αθεώρηση των τιμών. Εκεί θα έπρεπε να δίνουμε κάποια ευελιξία στους εθνικούς νομοθέτες. Να δούμε τώρα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ε, ταξιδιωτών και ειδικότερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε περίπτωση εκτάκτων ε, απρόβλεπτων ε, συνθήκων η οδηγία αναγνωρίζει στον καταναλωτή το δικαίωμα να ακυρώνει αν υπάρξει ε, ανωτέρα βία ή έκτακτες ε, ε, συνθήκες στον τόπο προορισμού και παρόλο που καταλαβαίνουμε την πρόταση θα θέλαμε να σας συμβουλεύσουμε να βασίσετε αυτό το δικαίωμα ακύρωσης σε επίσημους ε, συμβούλους ταξιδίων, κάτι το οποίο δεν θα δώσει πολύ μεγάλη ε, μεγάλο περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας. Όσον αφορά τον επαναπατρισμό σε περίπτωση εκτάκτων ε, συνθήκων, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε για παράδειγμα στην ιστορία, στην ομολογία του Γερμανικού Δικαστηρίου ότι το κόστος του επαναπατρασμού πρέπει τα δύο μέρη να το αναλαμβάνουν εξίσου. Ε, πρόκειται για παράδειγμα για την ε, νομολογία Τσέρνομπιλ, όπως την αποκαλούμε στη Γερμανία. Όταν πρέπει να γίνουν αποζημιώσεις ε, προς τον ε, καταναλωτή, 14 ημέρες προτείνει η οδηγία ως προθεσμία. Εμείς προτείνουμε ευθυγράμμιση της υποχρέωσης αυτής ε, με την υποχρέωση που συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία για τα δικαιώματα καταναλωτών που, αφορά, που αναφέρεται στην ε, αποζημίωση ε, του καταναλωτή χωρίς άχρηστες καθυστερήσεις. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο ενός τομέα που μερικές φορές οι συναλλαγές παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο μέχρι να λάβουν χώρα. Σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν από προηγούμενους ομιλητές, εμείς πιστεύουμε ότι η ευθύνη για τη σωστή τήρηση ενός ε, συμβουλέου βαρύνει τον ε, οργανωτή. Αν κάποιος ε, πουλάει κάποιες υπηρεσίες ως λιανοπολιτής και ως σύνολο της πουλά αυτές τις υπηρεσίες, θεωρείται οργανωτής. Οι λιανοπολιτές βέβαια είναι υπεύθυνοι για τα σφάλματα κρατήσεων και για τις πληροφορίες που ε, δίνουν στους καταναλωτές τους και πρέπει να έχουν συνυπευθυνότητα όταν πρόκειται για ε, οτιδήποτε πληροφορία λαμβάνει η χώρα πριν τη σύναψη μιας σύμβασης. Όσον αφορά τώρα την προστασία σε περίπτωση αφαιρεγιότητας, εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι οργανωτές, οι έμποροι πρέπει να δίνουν ένα αλφα επίπεδο προστασίας κατά της αφαιρεγιότητας, όπως επίσης και οι αεροπορικές εταιρείες. Διασυνοριακές πωλήσει πρέπει να καλύπτονται και οι ε, προμηθευτές πρέπει επίσης να προτείνουν μία ασφάλεια, κάτι το οποίο πρέπει να συμβαίνει βέβαια και σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς, Επίσης, ε, οργανωτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή υπάρχουν πολλές πωλήσει πλέον ε, από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που πολλούν τις υπηρεσίες τους στην Ευρώπη, πρέπει και αυτοί να καλύπτονται. Θα ήθελα να σας ζητήσω να δείτε τον κατάλογο των συστάσεών μας, ε, ο οποίος ε, είναι διαθέσιμος στο βάθος της αίθουσας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η κυρία Πέτρα Χάινικε θα είναι η επόμενη ομιλήτριά μας. Ε, Λειτουργεί το μηχάνημα. Μάλιστα. Καλό σας απόγευμα. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτό το θέμα σήμερα ενώπιον σας. Έχω γνωμοδότηση του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου στην Επιτροπή Αστικού Δικαίου. Έχω εργαστεί και εγώ για την εκπόνηση και για το αποτέλεσμα και το πόρισμα. Ε, θέλω να σας πω λίγο το background μου. Ε, στην επαγγελματική μου δραστηριότητα έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το δίκαιο τουρισμού. Ε, εδώ και 26 χρόνια εκπροσωπώ tour operators και πράκτορες σε ένα ευρύτατο φάσμα. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό, το είπε και ο κύριος Μάιερ. δεν ε, συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το θέμα των αεροπορικών εταιριών και των ταξιδίων. Θέλω να τονίσω ότι και το παραδοσιακό οργανωμένο ταξίδι, τα πακέτα δηλαδή, είναι πάρα πολύ προήρπτωκη υπόθεση. Είναι πολύ ενεχόμενη και αντισυμβαλόμενη και τα συμφέροντα. Αλλά όταν μιλάς για ένα οργανωμένο ταξίδι, για ένα πακέτο ας πούμε ταξιδιωτικό, υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα που μπορούν να ε, συνδυαστούν μέσα σε αυτό να κρύβονται από πίσω. Που εκ πρώτης όψεως δεν έχετε επίγνωση ας πούμε. Ε, οργανωμένα ταξίδια θεωρούμε ας πούμε ένα πακέτο, πετάς σε μια χώρα, πηγαίνεις ε, δύο εβδομάδες στη θάλασσα και ξαναγυρνάς. Υπάρχουν όμως ταξίδια κυνηγατικά, σαφάρι, περιπέτειας, εκπαιδευτικά, ανταλλαγή μαθητών που είναι και οργανωμένο πακέτο στο μεταξύ. Ε, όλα αυτά τα ταξίδια έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, τα προβλήματά τους και ε, τα χαρακτηριστικά τους. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι ένα απλό προϊόν αυτό που μας απασχολεί του οργανωμένου ταξιδιού. Είναι εξαιρετική η περιπλοκότητα και εδώ και 26 χρόνια δραστηριοποιούμε σε αυτό τον κλάδο και κάθε χρόνο έχω μια περίπτωση που λέω «Α, αυτό δεν το έχω ξαναδεί». Είναι τελείως καινούριο. Οι στόχοι της οδηγίας είναι αφενός η προστασία των καταναλωτών και αφετέρου η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού γέννη. Ε, θα αναρωτηθείτε ίσως τι δουλειά έχει εδώ στην προστασία των καταναλωτών εκπρόσωπος των διοργανωτών. Θα φανταστείτε ότι ε, είναι σε δεύτερη μοίρα για μας η προστασία των καταναλωτών. Δεν το πιστεύω. Γιατί και οι tour operators και οι πράκτορες ένα στόχο έχουν. Ε, τους ικανοποιημένους πολίτες και πελάτες να του φέρουν σόου ε, και αυλαβεί πίσω στο σπίτι τους. Και επίσης να είναι καλή η πληροφόρηση και ο πελάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται και να θεωρεί ότι του συμπεριφέρονται σωστά. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι και το ρόλο μου είναι ε, προκεχωρημένο φυλάκιο, ας πούμε, της υπηρεσίας εξυπηρέτησης των πελατών, γιατί έτσι το βλέπω. Ε, βεβαίως, ε, ε, είμαι και υπέρ της προστασίας των καταναλωτών, για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι ισόρροπη η πρόταση. Η ανταγωνιστικότητα στο διασυνοριακό εμπόριο και τουρισμό είναι βεβαίως ένα σημαντικό στόχο της οδηγίας, γιατί πράγματι είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες στην πρόσβαση στη γερμανική αγορά, ας πούμε, οι ξένοι tour operators ε, εκπλήσονται πάρα πολύ όταν βλέπουν τι κανόνες στη Γερμανία και πόσο διαφορετική είναι. Γενικά τώρα για την οδηγία. Πριν ρυθμίσει κανείς κάτι, καλό θα ήταν να το γνωρίζει. Δηλαδή ποια είναι η πρώτερη κείμενη νομοθεσία για να καταλάβουμε τι αλλαγές χρειάζεται και να ορίζουμε ξεκάθαρα κάθε φορά τι κάνουμε με σαφή περιχαράκωση και όρια και να αναρωτηθούμε αν η ρύθμιση την οποία προτείνουμε ανταποκρίνεται στους στόχους με ισορροπία και δικαιοσύνη προς όλους. Αυτό για την οδηγία μπορώ να το πω μόνο με κάποια παραδείγματα και σε πολλά σημεία χωλαίνει η κατάσταση και χωράει κριτική. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε από πού ερχόμαστε, ποια είναι η κείμενη νομοθεσία και ποια είναι τα ισχύοντα. Στην εισαγωγή της οδηγίας αυτό μεταφέρεται λανθασμένα. Λέγει ότι οι tour operators και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν την αστική ευθύνη για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα το βρείτε στο 1.1 παράγραφος 3. Αυτό είναι λάθος ε, ως διατύπωση στην οδηγία, ε, ως ισχυρισμός. Στην ισχύουσα οδηγία ε, την αστική ευθύνη έχουν οι πράκτορες όταν είναι αντισυμβαλόμενα μέρη. Οι απλοί, ε, τα πραπρακτορία δεν έχουν ε, αστική ευθύνη. Στη Γερμανία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στην Πορτογαλία βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα σε άλλα κράτη-μέλη. Το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έχει ευθύνη. Ε, δεν έχει παρουσιαστεί λοιπόν σωστά στην πρόταση για τη νέα οδηγία η κατάσταση που ισχύει. Το είπε και η κυρία Γκογιένς. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ορισμοί και σαφείς διαχωρισμοί που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στο άρθρο 3 ας πούμε, αν δείτε το πεδίο που καλύπτει το 2β Φερρυπίν. Και 2β πρώτο υποεδάφιο. Αν θέλετε λοιπόν να το ξεχωρίσετε από το 5α, τότε θα διαπιστώσετε ότι κάτι που είναι ενιαία διαδικασία κράτησης, τελικά να χρειάζεται πολλές συμβάσεις. Μπορεί ας πούμε ένα ταξίδι οργανωμένο να μην ε, εμπίπτει ε, στη συνολική αποζημίωση ε, ή να μην καλύπτεται για την περίπτωση της αφαιρεγκαιότητας. Μα η οδηγία θέλει να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να βοηθήσει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους tour operators να λειτουργούν διασυνοριακά με σαφείς κανόνες. Ε, δεν γίνεται αυτό με συγκεχημένους ορισμούς. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στους ορισμούς μας. Για τις ρυθμίσεις τώρα. Κάποιος προλαλή σας, νομίζω ο κύριος, είπε ότι η Ευρώπη δεν είναι νήσος. Όντως. Και στην οδηγία αυτή λέγεται ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών. Ισχύει αυτό. Τώρα, όταν έχει ένα ξένο tour operator που εδρεύει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα Ευρωπαίο ταξιδιωτικό πράκτορα, Ποιο θα φέρει την ευθύνη. Πώς θα ρυθμιστεί αυτό. Και για ποιο λόγο θα πρέπει να έχει ο εγχώριο πράκτορ την ευθύνη του tour operator. 71% των πελατών το 2011 είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και όλο και περισσότερο ο κόσμος κλείνει τα ταξίδια του από το διαδίκτυο και όλο και λιγότερο από ταξιδιωτικά πρακτορία. Έχει αλλάξει συμπεριφορά. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο πράκτορας, αλλά ένα tour operator είναι εκτός της Ένωσης, ποιος φέρει την ευθύνη. Εκείνος. Ε, ε, δεν είναι ελκυστικό το πακέτο αυτό και μπορεί κανείς να μην το κάνει πια και θα ε, χαθεί αυτό το μερίδιο αγοράς οι ε, πελάτες ε, θα ε, ψάχνουν στο διαδίκτυο τον Αμερικανό tour operator και θα αγοράζουν τα ταξίδια τους στο εξωτερικό εκτός Ευρώπης. Και πολλά από αυτά τα οργανωμένα ταξίδια έχουν πολύ επικίνδυνες δραστηριότητες. Παράδειγμα, φυσικά πάρκα, σαφάρι και τα λοιπά. Όλες αυτά τα ταξίδια περιπέτειας ε, ε, διεξάγονται πολύ ε, εκτός Ευρώπης και από οργανωτές εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, πάει ο καταναλωτής στο διαδίκτυο, αγοράζει το ταξίδι του από έναν τρίτο εκτός Ευρώπης του operator και προστατεύεται λιγότερο. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο στόχος της οδηγίας, μήπως να το σκεφτούμε και αυτό έτσι ε, και αντικειμενικά. Τώρα, για την ε, ισορροπία και την αποζημίωση, την δίκαιη, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην οδηγία και πάλι υπάρχει μια νέα ρύθμιση για το δικαίωμα αύξησης των τιμών. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο διοργανωτής να αλλάζει την τιμή, να υπάρχει μια τέτοια επιφύλαξη στη σύμβαση, με βάση πολύ περιορισμένα κριτήρια, να αλλάξει το ταξίδι, την τιμή, ε, αλλά η αύξηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, λέει, το 10%. Μέχρι εδώ καλά. Αυτό ακούγεται λογικό εκ πρώτης όψεως. Ο διοργανητής όμως του ταξιδιού θα πρέπει στο μέλλον να έχει τη δυνατότητα να κάνει εκτόσεις και προσφορές. Προς τα κάτω δεν έχουμε περιορισμό. Θέλουμε, λέει, να μειωθεί η γραφειοκρατία. Τι θα συμβεί εάν κάθε ταξιδιώτης έχει την αξίωση όταν μειώνονται ας πούμε, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες να φτηνένει και το πακέτο. Θα πρέπει να επανυπολογίσει ο διοργανωτής. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πότε κλείνει το ταξίδι, την ημερομηνία και την ώρα. Και ε, από τη στιγμή που αγοράζεις το πακέτο μέχρι που θα ταξιδέψεις, Μπορεί αν το γκρουπ είναι 20 άτομα να <laughs> χρειάζεται να κάνει 20 διαφορετικούς υπολογισμούς με βάση την ισοτιμία και ο καθένας να πληρώνει κάτι άλλο να είναι επιστροφή ενός ευρώ για τον καθένα. Με τεράστια γραφειοκρατία. Νομίζω θα πρέπει να βάλουμε ένα κατώτατο όριο εδώ που μπορεί να ισχύει και για τις δύο πλευρές. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί έτσι και αλλιώς θα πρέπει να συνυπολογίσουμε στον υπολογισμό ένα παράγοντα ε, αβεβαιότητας. Δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα. Δεν θα υπάρξει οργανωμένο ταξίδι που να μην αλλάξει κάποια μεταβλητή, ε, κάποιους παράγων που συνυπολογίζεται στον τιμολόγηση και στο κόστος. Και θα ήταν εξωφρενικό κάθε φορά να μπορεί και να υποχρεούται ο διοργανωτής να μειώνει την τιμή προς τα κάτω όταν έχει επιφυλαχθεί να προσαρμόσει την τιμή. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή τη ρήτρα διοργανωτής. Αλλά δεν το γράφει η οδηγία. Του λένε μπορείς να το αυξήσεις το πολύ μέχρι 10%. Τι συμβαίνει όμως εάν οι συναλλαγματικές οτιμίες αλλάξουν δραματικά ή διπλασιαστούν τα έξοδα καυσίμου και κάποια άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο 8β εάν υπάρξουν ριζικές μεταφορέ. Εγώ που είμαι ο tour operator και έχω το κόστος μου να τριπλασιάζεται, τι θα κάνω. Δεν μπορώ να το μετακυλήσω στον πελάτη. Αυτός ο κανένας νομίζω έχει αποφασιστεί επιπόλαια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν υπερβαίνει ένα ποσοστό η αύξηση, έτσι λέει η κατάσταση στη Γερμανία, μπορεί ο πελάτης να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει αποζημίωση. Αυτή είναι μια λύση κατά την άποψή μου λογική ε, σε αντίθεση με αυτή που προτείνεται εδώ, με αλφαγιώτα. Μάλλον, και μάλλον σίγουρα έχω εξαντλήσει το δεκάλεπτό μου. Είναι πολλά τα προβλήματα, μόνο ακροθυγός μπορώ να σας τα αναφέρω. Η βασική στόχη, ιδιαίτερα η ελάφρυνση και η διευκόλυνση του διασυνοριακού τουρισμού και η καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των Ευρωπαίων tour ε, operator είναι κάτι που μας χαροποιεί. Αλλά η προστασία των καταναλωτών δεν είναι προφανής από την οδηγία αυτή, γιατί για μένα ως Γερμανίδα πολλά πράγματα ε, είναι αυτονόητα. Όταν γίνει ένα λάθος στην κράτηση βεβαίως ε, είναι υπέτειος ο πράκτορας. Ή στο click-through ε, υπάρχει ένα θέμα του περικητήριου εφαρμογής. Α, κάτι άλλο που ήθελα να σας αναφέρω, Το τελευταίο. Θέλετε, λέτε, να προστατεύσετε τους καταναλωτές, να είναι πιο απλά τα πράγματα για τον καταναλωτή και όχι πιο δύσκολα, αλλά στο άρθρο 2 εξαιρούνται τα οργανωμένα ταξίδια, τα πακέτα στο 2 δέλτα, 2-2 δέλτα, D, και λέει στο 3-1 αλφαβήτα ορίζεται η ταξιδιωτική υπηρεσία και καθώς επίσης και μια περαιτέρω υπηρεσία σύμφωνα με το ΔΕΛΤΑ που είναι λοιπές τουριστικές υπηρεσίες που δεν θεωρούνται δευτερεύουσες για ε, μεταφορά ταξιδιωτών, ε, διανυκτερεύσεις, ενοικίαση αυτοκινήτων και κάτι αντίστοιχο. Ακόμα και αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες για να χαρακτηριστούν τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού εάν δεν είναι σημαντικό ποσοστό του οργανωμένου ταξιδιού, εξαιρείται από την οδηγία. Καλώ τα προβλήματα. Γιατί τι θα πει σημαντικό ε, ποσοστό του ταξιδιού. Είναι σημαντικό όταν κοστίζει πάρα πολύ. Ας πούμε, κλείνω ένα ταξίδι στο Αμβούργο ε, και θέλω να πάω να δω ένα musical. Όταν είναι 10 ευρώ το ειστήριο του musical, είναι σημαντικό τμήμα ή όχι είναι σημαντικό τμήμα το musical, γιατί γι' αυτό μπορεί να έχω πάει στο Αμβούργο, μόνο και μόνο για να πάω ε, να δω αυτή την παράσταση. Είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό, το σημαντικό πώς ορίζεται. Όλα αυτά είναι ασαφή και ε, παντού υπάρχει στην οδηγία αυτή η χρήση ε, κατάλληλα, δέοντα, αρμόζοντα σημαντικά. Τα ξέρω από την εμπειρία μου ότι ασάφειες δημιουργούν και μόνο και προβλήματα και τελείνουν τα προβλήματα ε, που θέλουμε να λύσουμε την οδηγία αυτή. Συμφωνώ με την κυρία Γκόγιενς, δεν χρειάζεται να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις και θέλω να το πω κι εγώ, ε, οπωσδήποτε να μην βιαστούμε. Το δίκαιο για τα αργονομένα ταξίδια αξίζει μια σωστή ρύθμιση. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουμε και πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε ολόκληρο το ταξίδι, όπως είπε η κυρία Γκόγενς, εκεί έχω μεγάλες επιφυλάξεις. Αλλά ε, και μόνο τα αργονομένα ταξίδια, τα πακέτα δηλαδή, ε, είναι μια ε, περίπλοκη παροχή υπηρεσιών και οι διακοπές των πελατών είναι περίπλοκα πράγματα και έχουν το δικαίωμα να περνούν τις διακοπές τους σωστά και με ασφάλεια. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Κρίστοφ Κλένερ, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής ε, υπηρεσίας ε, τεχνολογίας και υπηρεσιών ε, και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δω αν δουλεύει αυτό το σύστημα. δουλεύει. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ όλους, όλη την ανεξάρτητη ταξιδιωτική βιομηχανία και όλους τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Θα ήθελα ίσως να διορθώσω μία λανθασμένη εντύπωση που κυκλοφορεί ότι όλοι οι πράκτορες ε, είναι καμικάζοι. Λειτουργούν τη νύχτα, έρχονται, σου προσφέρουν μια υπηρεσία και δεν ε, σέβονται καμία νομοθεσία. Εγώ θα έλεγα ότι εκπροσωπώ εταιρείες Ε, εκπροσωπώ εταιρείε σοβαρές που λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς ε, θεωρούμε ότι το περιεχόμενο της οδηγίας είναι αυτονόητο. Ε, είναι οι απαιτήσει των καταναλωτών, θα πρέπει να, τους, έχουμε τους καταναλωτές ικανοποιημένους, άρα θα το εφαρμόσουμε. Αναγνωρίζετε κάποιες, σίγουρα όλες αυτές τις εταιρείες που εκπροσωπώ είναι κάποιες εταιρείες που ανήκουν ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι από τις Ηνωμένε Πολιτείε, κάποιες ευρωπαϊκές, είναι, λειτουργούν στα πλαίσια μιας ενιαίας αγοράς, ε, ούτως ή άλλως ε, το να καταργηθούν τα σύνορα και τα εμπόδια στην, στα ταξίδια είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Πιστεύουμε ότι το κείμενο της Κομισιόν έχει πολλά, πολλά, κάποια σημεία πάρα, πολλά, πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, διορθωθούν και το Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα να διορθώσει τα πράγματα. Και όπως είπε και ο κύριος Μάγερ, θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών με μια ενιαία και ανοιχτή αγορά. Προφανώς συμφωνώ και εγώ ότι δεν χρειάζεται να βιαστούμε να περάσει η νομοθεσία. Είναι καλύτερα όταν προσπαθείς ε, να ρυθμίσεις μια δυναμική αγορά, να τα σκεφτείς τα πράγματα καλύτερα και να ασχοληθείς με θέματα αρχής και όχι να μεταφέρεις κάποια ε, επιχειρηματικά μοντέλα σε, και να προσπαθήσει να τα προσαρμόσει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο 20-30 ετών. Τώρα, θα ήθελα να ασχοληθώ με τις ε, ιδιαιτερότητες του, της online business. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε προστασία του καταναλωτή καταρχάς, αλλά και ε, προσαρμογή στις ε, εξατομικευμένες ε, ανάγκες του καταναλωτή. Ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ο καταναλωτής έχει τώρα δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Το ένα είναι το δικαίωμα επιλογής και το δεύτερο χαμηλότερες τιμές επιλογή διότι μια δυναμική online αγορά σου επιτρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε πολύ περισσότερες εναλλακτικέ λύσεις από ό,τι στο παρελθόν και η τιμή ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν μεγάλοι online πολιτές που μπορούν να διαπαραγματευτούν πολύ καλύτερες τιμές, ε, χονδρικά αν θέλετε, από τους ε, πάροχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό ε, επιτρέψαμε σε πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη να ταξιδεύουν πολύ πιο συχνά. Και μέσα στα πλαίσια τη νομοθεσία αυτή, θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Δηλαδή θέλουμε μια νομοθεσία η οποία θα επιτρέπει να συνεχίσει η άνθηση αυτής της βιομηχανία ή θα βάλουμε κάποια εμπόδια και θα ε, διακινδυνεύσουμε τον περιορισμό τη ε, της δυνατότητας επιλογής που έχει ο καταναλωτής και να αυξήσουμε και το κόστος. Πιστεύουμε επίσης, όπως είπα και νωρίτερα, η... Η... ταξιδιωτικά γραφεία, τα ταξιδιωτικά πρακτορία online Έχουμε συμφωνήσει τα δυναμικά πακέτα που πουλάμε να καλύπτονται από, αυτόν τον, από αυτήν την νομοθεσία για να υπάρχει μια ομοιόμορφη αγορά. Αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στην νομοθεσία, να υπάρχει νομική σαφήνεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Όμως πιστεύουμε ότι αν διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας και ιδίω όσον αφορά ε, η, τις συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, διότι θα υπάρχει μια ενδεχόμενο τρέβλωσης κυρίως ε, όσον αφορά την ερμηνεία που θα δίνει το κάθε κράτος μέλος, αλλά και γιατί αυτή η νομοθεσία που έχουμε τώρα κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί και την επόμενη μέρα κάποιος θα ε, εφεύρει ε, ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα ξεφεύγει από το, από το δίκτυο, αν θέλετε, του διαδικτύου. Θα ξεφύγει από το διαδίκτυο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχω εδώ, έχουμε εδώ πέρα ε, τους φίλους μας από την ΑΙΑΤΑ και τις ε, αεροπορικές εταιρείες που δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος ελέφαντας αυτήν την αίθουσα. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι Υπάρχουν εταιρείες μεγάλες ε, ε, που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. και καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία, ενώ υπάρχουν άλλες, άλλες εταιρείε, άλλες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν και που δεν καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία. Έχουμε, να κάνουμε, έχουμε κάνει και κάποιες προτάσεις ε, στο κείμενο, σε ένα κείμενο το οποίο θα διανεμηθεί σύντομα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ενισχυμένη προστασία για τους καταναλωτές όταν ταξιδεύουν, αλλά το πρόβλημα είναι, είναι αυτή η κατάλληλη νομοθεσία για να συμβεί κάτι τέτοιο. Εδώ θέλαμε να, ρυθμίσουμε μια τελεία διαφορετική αγορά στο τέλος δεκαετίας του 80 και του 90 και αυτή η νομοθεσία μπορεί να ε, προστατεύσει τον τόσο προχωρημένο αν θέλετε χώρο ταξιδιού, ταξιδιού όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα ή να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή, να συμπεριλάβουμε τα δυναμικά πακέτα, κάτι με το οποίο συμφωνούμε, και μετά να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε σαν θέμα αρχής όλους τους ταξιδιώτε ε, ταξιδιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα ε, αν, αν έχουν κάνει μια κράτηση για εισιτήριο μόνο, για συνδυασμό υπηρεσιών κτλ. κτλ. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έτσι όπως είναι τώρα το πακέτο, θεωρούμε ότι είναι κάπως αυθαίρετη η κατάσταση. Λοιπόν, όταν μιλάμε για το πακέτο, να μιλάμε για συνδυασμούς που πολλούνται σε μία συναλλαγή και υπάρχει μία ενιαία τιμή, διότι όταν υπάρχει μία ενιαία τιμή, τότε είναι ένα πακέτο. Αυτός είναι ο ορισμός του πακέτου το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Όπως επίσης ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις διατάξεις που, ασχολούνται, που αφορούν τις συνδυασμένε αξιωτικές υπηρεσίες, διότι πιστεύουμε ότι αυτός δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δημιουργηθούν ε, συγχύσεις, ε, θα υπάρξει ενδεχόμενα στρέβλωση του αμυγονισμού και μια ενδυνάμει εκμετάλλευση από τις διάφορες εταιρείε που λένε ναι εντάξει εμείς ξέρουμε τους κανόνες και θα προσπαθήσουμε να τους παρακάμψουμε, ναι και τους γνωρίζουμε πλέον. Επίσης συμφωνώ με την Μισελ ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις εξαιρέσεις για, το, για τα επαγγελματικά ταξίδια, διότι εκεί υπάρχει ε, μια συγκεκριμένη σύμβαση ανάμεσα στις εταιρείες ε, και, στις, ε, και, στους, και στα ταξιδιωτικά γραφεία. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε την σχέση ανάμεσα στα συνδυασμένες ταξιωτικές υπηρεσίες και, την, και τα δικαιώματα του πελάτη. Ας πούμε ότι κάποιος έχει οργανώσει ένα ταξίδι, ε, έχει ακυρωθεί μια πτήση και ο επιβάτης δεν ταξιδέψει καθόλου και δεν ζητάει τίποτα από, τον, ε, από το ταξιδιωτικό γραφείο. Άρα δεν παίρνει αποζημίωση. Εδώ δημιουργείται μια σύγχυση και αυτό μπορεί να... Ε, θα μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές, επειδή δεν γνωρίζουν απόλυτα την νομοθεσία, να χάσουν κάποια χρήματα. Ε, γιατί, ας πούμε, αποφάσισαν να μην ε, ξεκινήσουν το ταξίδι και δεν ζήτησαν από τον πράκτορα να τους βρει μια εναλλακτική λύση. Επίσης, ε, τα επίπεδα προστασίας από την χρεοκοπία θα πρέπει να ε, υπόκεινται στον πραγματικό κίνδυνο. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα καταποκοπή ποσό. Ας πούμε, αν πάρετε το παράδειγμα της Expedia, που μπορεί να το ξέρετε. Όταν κλείσετε ένα, μια πτήση και ένα ξενοδοχείο με την Expedia, με τις περισσότερες... Ε, ε, στις η Expedia δεν βλέπει τα χρήματά σας τα χρήματα πηγαίνουν κατευθείαν στο ξενοδοχείο τουλάχιστον όσον αφορά το ξενοδοχείο και κατευθείαν στην αεροπορική εταιρεία ενδεχόμενα σεβόμενοι και τις προθεσμίες που βλέπει η ΑΙΑΤΑ. Αλλά συνήθως πηγαίνει κυρίως στους, ε, στους πάροχους των υπηρεσιών. Ε, άρα η, η, η χρεοκοπία της, η χρεοκοπία της, ε, του πράκτορα δεν παίζει κανέναν ρόλο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με, την ίδια, με τον ίδιο τρόπο ε, αυτή η περίπτωση με την περίπτωση όπου η εταιρεία έχει τα χρήματά σου από την αρχή μέχρι το τέλος και τα κρατάει. Επίσης, οι διασυνοριακές, ε, ε, οι εταιρείες που δρούν διασυνοριακά τέλος πάντων, δημιουργούν δημιουργείται στην περίπτωση αυτή κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τις εθνικές επιλογές. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, αν θέλετε, της συνεδρίασής μας, που αφορά τις ε, ερωτήσεις ε, που θα θέλαν να θέσουν οι συνάδελφοι. Τόνι εσύ έχει δει στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, επεξηγήσεις. Εγώ δούλεψα για ε, λίγα χρόνια στην ε, οδηγία για την χρονομεριστική μίσθωση, το timeshare. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελα να την αλλάξω αυτήν. Το μόνο που ακούω τώρα είναι παράπονα ότι πρέπει μια, να έχουμε μια εναρμονισμένη οδηγία. Μιλάμε όμως για την ευρωπαϊκή αγορά. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να έχουμε ισότιμη μεταχείριση ε, σε όλο το κλάδο, αλλά και το ίδιο επίπεδο προστασίας για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, δεν χρειαζόμαστε καταναλωτές. Ε, κανονισμό, συγγνώμη είναι ένα ελάχιστο πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να λύσουμε. Γιατί αν τα προβλήματα είναι σε εθνικό επίπεδο, τότε οι διάφορες επιχειρήσεις θα διαλέξουν τις χώρες ανάλογα με την ομοθεσία που έχουν αυτές και οι υπόλοιπε δεν έχουν ε, τη δυνατότητα ισότιμης μεταχείρισης δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία, ούτε για τους καταναλωτές, ούτε για τον ε, κλάδο αναψυχής. Εσείς θα προτιμούσατε οδηγία ή κανονισμό, ρωτάω εγώ τους προσκεκλημένους μας. Ευχαριστώ. Θα μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις και μετά θα δοθούν ε, οι απαντήσεις στο τέλος. Η κυρία Ριούλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μαζεψουμε ολες τις ερωτησεις και μετα θα δοθουν οι απαντησεις στο τελος κυρια ριουλε ευχαριστω πολυ θα ηθελα να επανέλθω σε ένα πρόβλημα που για μένα δεν έχει λυθεί, το πεδίο εφαρμογή. Αν κατάλαβα καλά, δεν το είπατε, αλλά το γράφει η παρουσίασή σας, είστε και υπέρ της ένταξης και των εξατομικευμένων ε, ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω πρακτορείων. Ναι, και θέλω να μιλήσω και σε σχέση με τον προλαλήσα, τον τελευταίο μιλητή. Οι νέοι όταν κάνουν κρατήσεις ε, για ένα ταξίδι θέλουν να έχουν την επιλογή να το οργανώνουν μόνοι τους το ταξίδι και τα διάφορα στοιχεία να τα συνενώνουν, να το οργανώνουν. Υπάρχει και ένα ρίσκο εκεί αλλά ταυτόχρονα και πιο φθηνές τιμές και τα δύο μαζί συνδυάζονται. Λοιπόν, τώρα αν ε, και σε περίπτωση που ε, εμπίπτει στην οδηγία και θα με ενδιαφέρει η απόψή σας, πώς πρέπει να γίνει αυτό και πώς θα την κάνουμε ε, δελεαστική όλη αυτή την πρόταση για τους νέους χρήστες. Uh, so I think next is uh, Mrs. McClarkin. Uh, thank you, Chairman, and thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους Συγγνώμη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το όνομα του τελευταίου ομιλητή. Πάντω, ε, ανέφερε το θέμα τη τιμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για του καταναλωτέ. Μα ενδιαφέρει πολύ το προστασ... η προστασία των καταναλωτών, αλλά έχει και ένα τίμημα. Και δεν άκουσα για τους... από του υπόλοιπου ομιλητέ ποιο ακριβώ θα το πληρώσει αυτό το τίμημα. Και είστε, ότι, είστε ε, εκπρόσωποι των οργανώσεων καταναλωτών και λέτε ότι δεν έχουν πρόβλημα οι καταναλωτέ να πληρώσουν το τίμημα. Ε, όταν εγώ ταξιδεύω και το κάνω συχνά, μου αρέσει το γεγονός ότι έχω την επιλογή, μπορώ να, να, μπορώ να τα διαλέξω όλα μόνη μου και να δημιουργήσω το δικό μου πακέτο online. Το αποδέχομαι ότι ε, είναι ε, ένας τρόπος να μειώσω το κόστος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το κόστος για τους καταναλωτές. Πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό ώστε από τη μία να υπάρχει επίπεδο προστασίας και από την άλλη να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν πακέτα ε, προσιτών τιμών. Thank you. Um, I think is next on my list. Η κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία μικρή παρέμβαση Βλέπω στο κείμενο αυτό, καταρχάς κάποιος είπε, νομίζω ο τελευταίος ομιλητής, ε, ότι πρέπει να συνδεθούν τα δύο κείμενα και το κείμενο των ε, δικαιωμάτων ε, των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Εγώ είμαι η, συγητή, η της Επιτροπής Μεταφορών για το θέμα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ε, δεκάδες διαφορετικούς ορισμούς σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Συζητάμε τόσο πολύ για τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Ε, πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση και για τα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και το, τις αποζημιώσεις. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την οδηγία και αυτό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον κοινή ευθύνη μεταξύ του λιανοπολιτή και του, οργανωτή του ταξιδίου. Ε, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το δικαίωμα του καταναλωτή και μπορούμε πραγματικά να το αποδυναμώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, πιστεύω και συμφωνώ ε, με την κυρία Γκόγεν σε αυτό, ότι η πλήρης εναρμόνιση, ειδικότερα όταν μιλάμε για πλήρη εναρμόνιση λέμε ότι είναι τι ωραίο πράγμα αυτό, αλλά ξέρουμε καλά ότι στα ευρωπαϊκά κείμενα η πλήρης εναρμόνιση είναι συχνά κάτι το οποίο μειώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών, ε, συγκεκριμένα των επιβατών, των ταξιδιωτών, όλων των καταναλωτών, γιατί ακριβώς ε, η νομοθεσία αφορά κάθε φορά ένα επίπεδο ε, προστασίας μεγαλύτερο. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε και με άλλα κείμενα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με αυτό το κείμενο, αλλά να μην βιαστούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο πριν από το τέλος κοινοβουλευτικής μας θητείας, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο και για την οικονομία αλλά και για τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Ε, το να βιαστούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Φώστερ νομίζω, mm καλώς ήρθατε από την Επιτροπή Μεταφορών. Δουλεύουμε πολύ, συνεργαζόμαστε πολύ στενά για την πρόταση αυτή. Ναι, είμαι και σκιώδης συγγήτρια για τα δικαιώματα των επιβατών ε, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το ότι είχαμε μια κρόση για το θέμα αυτό και εμένα μου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχασα δυστυχώς τις εισαγωγικά σχόλια, αλλά άκουσα τους ομιλητές. Ως παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι όταν ε, υπάρχει κάτι για 20 χρόνια, είναι γεγονός ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να το εξετάσουμε, ...αλλά δηλαδή, δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Για να μπορέσει λοιπόν να λειτουργήσει κάτι πρακτικά, πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο επικουρικότητα σε σχέση με το ποιοι είναι οι κανόνες και κανονισμοί σε σχέση με τα, ε, με την προστασία των καταναλωτών όταν ε, κλείνουν τις διακοπές τους οτιδήποτε άλλο. Γιατί με την αρχική οδηγία ήταν σαφή τα πράγματα. Ο κόσμος πήγαινε σε ένα ταξιδιωτικό πράκτορα έκλεινε, έκανε κράτηση για το αεροπλάνο και για το ξενοδοχείο Είπατε όμως ότι έχετε κάποιες ανησυχίες, είναι ότι τώρα πάει κανείς στο διαδίκτυο, ε, πατάει διάφορα κουμπιά, από το ένα site πάει στο άλλο. Ε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Από τη μία λέτε, από την άλλη, από, τη μία Λέτε ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάει στον ταξιδιωτικό πράκτορα άμα δεν του αρέσει αυτό, όμως ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να υπάρχει ε, καν. Και δεν το κρίνω αυτό, απλώς λέω ότι είναι η πραγματικότητα. Είναι ότι υπάρχουν πλέον ε, τέτοιες προσφορές και διάφορες τιμές για οποιονδήποτε, μέχρι και το φοιτητή που θέλει να ταξιδέψει, είναι τεράστια επιλογή και φυσικά είμαστε σε ανταγωνισμό με τις επιχειρήσεις ε, τρίτων χωρών. Είναι εντελώ διαφορετικά τα πράγματα. Θα χαλαρώσουμε λοιπόν και να δούμε ε, ποιοι χειρίζονται τα θέματα αυτά εντό της Ευρώπης Πολλέ φορέ όμως οι ανταγωνιστές μας τρίτες χώρε δεν έχουν να συμμορφωθούν με κανέναν κανόνα και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σκέφτηκε λοιπόν πολύ διεξοδικά το θέμα. Δεν νομίζω ότι έχουν ακόμη τα, τις απαντήσεις και δεν νομίζω ότι υπήρξε επαρκή συζήτηση με τον κλάδο. Ε, για όλα αυτά τα θέματα, τα θέματα των ιστοτόπων για παράδειγμα Orbit και λοιπά τα οποία αναφέρατε δεν νομίζω ότι έχουμε όλα τα ερωτήματα, τα, τις απαντήσεις στα ερωτήματα, γιατί αν δούμε τα θέματα της αφαιρεγγιότητας, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε, για παράδειγμα, εάν ο Τζον πάει εδώ, ε, κλείσει μία πτήση, μετά πάει πιο πέρα και κλείσει ένα ε, ξενοδοχείο, αν κάτι πάει στραβά δεν ξέρει σε ποιον να απευθυνθεί. Πολύ καλά λοιπόν τα λέμε ως, προ προς την προστασία των καταναλωτών. Πολύ καλό είναι αυτό. Καλό είναι να υπάρχει και καλή εξυπηρέτηση πελετών. Αλλά πώς είναι να το προχωρήσουμε όταν δεν έχουμε λύσει τις απορίες μας. Και θα ε, ολοκληρώσω τώρα κύριε Πρόεδρε. Είναι ότι πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις αλλά να είναι και πρακτικέ. Δεν έχει νόημα να έχουμε λύσει που δεν θα προστατεύουν τον καταναλωτό, αλλά αντιθέτω υπονομεύουν την επιλογή που θέλουμε να του δώσουμε. Οπότε, καλή επιτυχία σα εύχομαι, αλλά πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Ήταν εξαιρετική ιδέα λοιπόν να έχουμε τη σημερινή ε, ακρόαση και σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε τη δυνατότητα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμεί, κυρία Φώστερ και ευχαριστώ όλου όσου πήραν το λόγο. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τους τέσσερις ε, εμπειρογνώμονές μας ε, σε μερικά λεπτά, έκαστος, ε, κατά τις πέντε πρέπει να ολοκληρώσουμε, να απαντήσετε. Και η κυρία Μανφρέντι, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλει να μας κάνει ορισμένα σχόλια. Και να δώσω και το λόγο και στον εισηγητή, τον κύριο Μάιερ. Αν συμφωνείτε λοιπόν, εντάξει, μπορεί να ξεπεράσουμε λίγο τις πέντε να αρχίσω λοιπόν με την Μονίκ Γκόινς και μετά με τους υπόλοιπους ομιλητές. Να σας καλωσορίσω κιόλα. Ε, είμαι βέβαιος ότι και ο αντιπρόεδρος μας το έκανε. Σχετικά με την πρόταση να έχουμε ένα κανονισμό και όχι οδηγία, Νομίζω ότι οι υπηρεσίε της Κομισιό ήδη έχουν αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση σε αυτή την τόσο περίεργη και περιπλοκή αγορά. Επομένω, το να μπερδέψουμε και την, τα πράγματα ζητώντας έναν κανονισμό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μιλάμε για συμβασιακό δίκαιο εδώ. Ε, επομένως, ε, είναι πολύ επικίνδυνο να προχωρήσουμε ε, σε μια τόσο απόλυτη και λεπτομερή ρύθμιση. Ε, δεν θεωρούμε ότι το κατάλληλο νομοθετικό όργανο είναι ούτε ο κανονισμός, ούτε μια λεπτομερής ε, ε, οδηγία πλήρους εναρμόνωση. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι η νομοθεσία που διέπει τους τομείς αυτούς δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Εντάξει, Θέλουμε να εξασφαλίσουμε το, το υψηλότερο βαθμό ε, προστασίας του καταναλωτή, αλλά θα πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Όπως είπε και Μισελ, να έχουμε μια εναρμόνιση κατά επιλογή, δηλαδή ε, ε στα σημεία όπου υπάρχει επαρκής προσέγγιση μπορούμε να έχουμε πλήρη εναρμόνιση. Σε άλλα σημεία όμως δεν μπορεί να γίνει όσον αφορά τις υπηρεσίες καταναλωτή, όντως ε, σε έναν ιδανικό κόσμο οι καταναλωτές και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ε, προστατεύονται από τον ίδιο τρόπο ανάλογα με τις υπηρεσίες που απαιτούν. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έτσι όπω έχουν τα πράγματα δημιουργείται μια σύγχυση στους καταναλωτές και χρειάζεται μια αναθεώρηση. Έτσι όπως ε, είναι τα πράγματα, δεν θέλουμε να προσθέσουμε και άλλο ένα επίπεδο περιπλοκότητας και σύγχυσης, διότι όπως είπε και η Κρίστα, θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση ε, για το πακέτο, για τις συνδυασμένες αξιωτικές υπηρεσίες. Ε, πρέπει να αυτοί οι ορισμοί να συμπεριληφθούν εδώ, δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως <laughs> όλος αυτός ο τομέας είναι ο παράδεισος των δικηγόρων. Υπάρχουν τόσες διατάξεις που πρέπει να εξηγηθούν και να διευκρινιστούν. Σχετικά με τις τιμές, κάθε στοιχείο προστασίας του καταναλωτή κοστίζει. Και συμβαίνει αυτό και για την ασφάλεια των τροφίμων και για, το, και για τα ταξίδια, για, τα, για τον ιατρικό εξοπλισμό, για τα φάρμακα κτλ. Στο πλαίσιο αυτό, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτό το οποίο σου προσφέρεται σαν ε, προστασία αντιστοιχεί στην, ε, στις προσδοκίες σου, στις νόμιμες προσδοκίες σου. Και ο καταναλωτής πρέπει να ε, προστατεύεται και έχει το δικαίωμα να απαιτήσει προστασία. Και δεν είναι μονάχα η χρεοκοπία ή η κακή παροχή υπηρεσιών. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε ότι δικαιούται, δικαιούται ο καταναλωτής προστασία. Δεν θα πρέπει λόγω μιας τεχνητής τεχνική, διάκρισης να βρεθεί ο καταναλωτής εκτός προστασίας. Και εδώ πρέπει να διευκριστεί το πράγμα. Και τώρα βέβαια, εάν είσαι, δικαι... Ε, ε, είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις το κίνδυνο, τότε θα πρέπει να έχεις και μία μείωση της τιμής τους. Της τιμής. Τώρα, όπως είπε και η κυρία Βανιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τοποθετήσεις την οδηγία στο σωστό της περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να εντοπίσουμε τις συνδέσμους που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτή την οδηγία και στα κείμενα, τα νομοθετικά κείμενα και νομοθετικές πράξεις που ήδη ισχύουν. Ο κύριος Ντεμπλούστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, καταρχάς, η ερωτήση του κυρίου Μάντελς. Πιστεύουμε ότι εμείς, ε, η βιομηχανία συμφωνεί με τους καταναλωτές στο σημείο αυτό. Ένας κανονισμός ε, θα περιπλέξει τα πράγματα και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να λύσει. Ε, εξαρτάται από την νομοθεσία των κρατών μελών Επίσης εξαρτάται και από την πρόσβαση στο επάγγελμα και οι διατάξεις πρόσβαση στο επάγγελμα του πράκτορα ή του οργανωτή και ε, ταξιδίων ε, διαφέρει από κράτος και σε κράτος, άρα θεωρούμε ότι ο κανονισμός τελικά δεν θα διευκολύνει ε, τον κλάδο. Εμείς όμως υποστηρίζουμε ένα υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης, ε, είναι η στοχευμένη εναρμόνιση όπως λέω στο κίνημά μου. Ενιαίες υπηρεσίες και σε σχέση με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες ε, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης από ό,τι θυμάμαι, δεν, υπήρχε, δεν υπήρξε κανένας ε, ενδιαφερόμενος ε, που να καλύπτει τις ενιαίες υπηρεσίες, που να θέλει να καλύπτουν τις ενιαίες υπηρεσίες ή εξατοδικημένες υπηρεσίες σε αυτή την οδηγία. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν οποιονδήποτε πράκτορα. Τους προσανατολίζει η τιμή. Μπορούν να επιλέξουν οποιονδήποτε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τους ενδιαφέρει, η τιμή, όταν κάνεις μια κράτηση, δεν είναι για ταξίδι, δεν είναι για διακοπές, ή οτιδήποτε άλλο, το, αποτελεσμα... το στοιχείο το αποφασιστικό για τα εκατομμύρια καταναλωτών στην Ευρώπη είναι η τιμή. Έχουμε θέσει το ερώτημα στην, ε, στην Κομισιόν πολλές φορές. Έχουμε ερωτήσει την κυρία Μανφρέντι πολλές φορές και άλλους συναδέλφους και έχουμε και έναν εξαιρετικό διάλογο με τις υπηρεσίες της Κομισιόν και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο καταναλωτής ε, αυτό το οποίο, το οποίο ενδιαφέρεται είναι η τιμή. Δεν είμαι σίγουρος ότι μας άκουσαν. Οι συμπληρωματικές υποχρεώσεις που έχουν ε, βέβαια προφανώς κοστίζουν και υποχρεώσεις σημαίνουν ε, συμπληρωματική ασφάλιση και στο τέλος είναι βέβαια να δούμε ποιος πληρώνει το καταναλωτή. Ο, ο καταναλωτής μπορεί να είναι σε ένα site ε, στην Κίνα, της Κίνας, της Αργεντινής κτλ. Και εκεί βρίσκει το ίδιο πακέτο 50 ευρώ ε, ευθυνότερα ανάτομο και είναι μια τετραμελής οικογένεια. Μπορείτε να φανταστείτε βέβαια από ποιον θα ψωνίσει ο καταναλωτής. Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό που, ε, τον, ανταγωνισμό σε, όλη την, σε όλο τον πλανήτη αν θέλετε και δεν θα πρέπει να, ε, το ξεχνάμε αυτό. Η, στην Ευρώπη βέβαια τα πράγματα είναι ε, κάπως πιο ε, απλά αν θέλετε. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι οι προτάσεις που γίνονται για τα οργανωμένα ταξίδια και για τις συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες πρέπει να είναι σαφής, να μην υπάρχουν επικαλύψεις, οι, οι, οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται είτε έχουν κλείσει ένα εισιτήριο μόνο είτε έχουν κλείσει ένα πακέτο. Επίσης σχετικά με τις παρατηρήσεις κυρίας Φώστερ για την ανάγκη να αλλάξουμε μια οδηγία που 25 ετών για την προστασία της ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου συμφωνώ απόλυτα, επομένως ε, μπορώ να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Χάνικε. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για την εναρμόνιση των δικαιωμάτων των ε, ε, πιβατών και σχέση με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Έχει νόημα συναφής υποθέσεις να ρυθμίζονται με νέο τρόπο ή με παρόμοιο τρόπο και να μην βάζεις ε, στο ένα όριο 3,5 ευρώ, στο άλλο 4 ευρώ. Το θέμα είναι ε, ο στόχος κάθε φορά, αν υπάρχει σωστή στόχευση και αν είναι κατάλληλη. Γιατί ένας καταναρωτής που αγοράζει μόνο το ταξίδι, την πτήση δηλαδή, ε, περιμένει ε, λιγότερη υποστήριξη από τον αερομεταφορέα από ότι εκείνο που αγοράζει ένα οργανωμένο ταξίδι, ένα πακέτο ε, και πάει κάτι στραβά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Δηλαδή όταν αγοράζεις ένα συνολικό πακέτο περιμένεις για μεγαλύτερη και διαφορετική προστασία. Όταν αγοράζεις ένα αεροπορικό στήριο και μόνο, αλλιώς βλέπεις τις ανάγκες προστασίας σου ε, ως καταναλωτή σε σχέση με τον πάροχο της υπηρεσίας. Ήταν σημαντικό να το πω αυτό. Κατά τα άλλα, η Ευρώπη δεν είναι νήσος, είπαμε, δεν είναι νησίδα κάπου. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο καταναλωτής στον δρόμο προς την πιο φτηνή τιμή ε, μπαίνει σε μονοπάτια και σε ατραπούς που δεν ε, του παρέχουν από καμία προστασία μέχρι πολύ χαμηλή ή χαμηλότερη από την ευρωπαϊκή. Και ο πράκτορας που προσφέρει ένα πακέτο ενό ξένου tour operator δεν θα γίνει ποτέ ο ίδιο tour operator. Δεν αναλαμβάνει τέτοια ευθύνη. Αν το κάνει είναι θεοπάλαβο. Διότι έχει ένα ε, ελάχιστο περιθώριο κέρδου και εκτίθεται σε ένα τεράστιο κίνδυνο. Θα πρέπει όμως να ενημερώνεται ο πελάτης για το ρίσκο που διατρέχει και αυτό έχει νόημα να το κάνει ο πράκτορας. Γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να καταλάβει και με τα λόγου γνώσεως ε, ο καταναλωτής να ξέρει σε τι κίνδυνο εκτίθεται και σε τι ε, ρίσκο μπορεί να πέσει. Από πού θα κλείσω και θα αγοράσω το ταξίδι. Από ένα Ευρωπαίο πράκτορα που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβό αλλά παρέχει μεγαλύτερη προστασία. Να είναι ελεύθερο στην επιλογή του. Βεβαίως κανείς δεν προστατεύεται παρά τη θέλησή του αλλά θα πρέπει να γνωρίζει τα επίπεδα αυτά και να τα αποφασίζει μόνος του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τον ενημερωμένο πολίτη και τον ενημερωμένο καταναλωτή που είναι και ένα στοιχείο της ελεύθερης επιλογής. Μπορεί ο άλλος να σου πει δεν με ενδιαφέρει η προστασία, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η φθηνή τιμή, αλλά να τα γνωρίζει όλα αυτά. Και την ενημέρωση μπορεί να την ανθέσει κανείς στον πράκτορα, όχι όμως και στην όλη την ευθύνη. Ευχαριστώ. Thank you, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το ερώτημα οδηγία ή κανονισμός ε, θα συμφωνήσω με την Μονίκ. Καλή τύχη αν θέλετε να το κάνετε κανονισμό αυτό. Εκπροσωπώντας βέβαια εταιρείες διακόπτει ο μιλητής, εκπροσωπώντας ε, οργανισμούς ε, που είναι από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όσο πιο μεγάλη εναρμόνιση υπάρχει, τόσο το καλύτερο. Αλλά να αρχίσουμε από απλά πράγματα, πρόσβαση στη, στα εθνικά προγράμματα προστασίας κατά της αφαιρεγγιότητας. Μερικές φορές η πρόσβαση αυτή περιορίζεται σε φορείς που έχουν την έδρα στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το, να το ρυθμίσουμε αυτό. Ίσως και να μπορούμε. Υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, που το καθιστούν ευκολότερο ε, για κάποιους ε, φορείς, για κάποιες εταιρείες να δραστηριοποιούνται και σε άλλες χώρες. υπάρχουν τομείς που είναι δύσκολοι ω προς την προστασία των καταναλωτών. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, αλλά μπορεί να φτάσουμε σε κάποια εναρμόνιση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συναλλαγέ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ερώτημα του πώς μπορεί η προστασία των καταναλωτών ε, να είναι πιο ελκυστική για τους νέους ε, σε σχέση με το κόστος της προστασίας Νομίζω ότι αυτό συνάδει με το δικό μας σκεπτικό. Όταν εξετάζουμε τους καταναλωτές μας και κάνουμε μεγάλες έρευνες για το τι ζητούν ε, οι καταναλωτές, προφανώς ο κάθε καταναλωτής είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές απαιτήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να κάνει μια διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών, τέλος πάντων μεταξύ δύο, ε, κατηγοριών με υποκατηγορίες. Υπάρχουν οι πελάτες που μπορούν να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Ε, από την πτήση μέχρι τη μετάβαση στο ξενοδοχείο θέλουν να τα καλύψουν όλα. Κάποιον να τους απαντήσει τις ερωτήσεις ε, τόπο ε, στο ξενοδοχείο που θα διαμείνουν, όλα τα πάντα, το φαγητό, τα ποτά, τα πάντα. Αυτό είναι ένα είδος καταναλωτή. Και αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Που όλο και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν τέτοιου είδους ε, ταξιδιωτική εμπειρία. Είμαι διατεθειμένος να το πληρώσω, να πληρώσω για αυτή την πλήρη προστασία. Υπάρχει όμως ε, και μια ομάδα η οποία ε, ταξιδεύει με πολύ λίγα μέσα και θέλει να έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Ε, πρέπει να τύχουν ε, εκμετάλλευσης. Όχι βέβαια. Κατά πόσο πρέπει να τους ενημερώνουμε για τις επιλογές ε, που έχουν ως προς το επίπεδο προστασίας τους. Ναι, βεβαίως πρέπει να τους ενημερώνουμε. Από τότε που είχαμε την πρώτη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας του 2009, είχαμε επιχειρηματολογήσει τότε ε, ότι θα έπρεπε να υπάρχει υποχρέωση από τους ταξιδιωτικούς, του ταξιδιωτικού πράκτορα να ενημερώνει ή να προσφέρει μια ασφάλεια, για παράδειγμα. Δεν είναι υποχρεωτικό για τον καταναλωτή να ασφαλιστεί, αλλά τέλος πάντων να είναι μια σαφής επιλογή σε σχέση με τη διαφανή πληροφορία που μπορεί να πάρει ο καταναλωτής. Και εντάξει, μπορούμε από εκεί πέρα να ρυθμίσουμε τι θα περιλαμβάνει αυτή η διάταξη περί ενημέρωσης. Κανένας λοιπόν δεν έχει από μόνος του τις απαντήσεις, αλλά ίσως μπορούμε να βρούμε τέλος πάντων κάποιες, κάποια, κάποιες ενότητες ε, που να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Αναφερθήκατε ε, στη σχέση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με των δικαιωμάτων των επιβατών. Προφανώς Προφανώς υπάρχουν σχέσεις, ε, υπάρχουν βέβαια και ορισμένα αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ της οδηγίας για τα οργανωμένα πακέτα και των ε, επιβατών αεροπορικών εταιριών και πρέπει να λυθούν γιατί μερικές φορές πολλοί καταναλωτές νομίζουν ότι έχουν πάρει σωστή απόφαση, φτάνουν στο αεροδρόμιο, έχουν μια ώρα να αποφασίσουν ε, που, τι θα κάνουν, μένω σπίτι, περιμένω την επόμενη ε, πτήση, έχει ένα Σαββατοκύριακο μόνο στη διάθεσή του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανείς την απόφαση, γιατί κανένας ε, δεν έχει στο μυαλό του όλες τις λεπτομέρειες όλων αυτών των οδηγιών τη στιγμή που πρέπει να πάρει την απόφαση. Έχουμε κάνει λοιπόν πολύ συγκεκριμένε συστάσεις ε, στη... στο έγγραφο δεσιό μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την ε, πολύτιμη συμβολή σας ε, σήμερα. Ε, την εκτιμούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς έχουμε λιγάκι καθυστερήσει, αλλά η κυρία Σενέλοβα είναι εδώ και έχουμε ακόμη ένα θέμα να εξετάσουμε. Θα ήθελα παρόλα αυτά να δώσω το λόγο στην κυρία Μανφρέντι, να την καλωσορίσω, γιατί ήταν πολύ διαθέσιμη και συνεργάστηκε πολύ με το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Να σας δώσω λοιπόν λίγα λεπτά να μας ε, πείτε κάποια πράγματα και να δώσω και τη δυνατότητα στον Hans Peter Mayer να συνοψίσει τη συζήτηση. Κύριε Μανφρέντη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την οργάνωση αυτής της ακρόασης που δείχνει πραγματικά σε όλους μας ε, ε, πόσα ε, συμφέροντα υπάρχουν πριν πίσω από την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη μία καταλαβαίνω κάποιες επικρίσεις, από την άλλη βγαίνω από την αίθουσα αυτή πιστεύοντας ότι είναι μια εξισορροπημένη πρόταση αυτή που υποβάλαμε και είμαι σίγουρη ότι με τη βοήθεια τη δική σας και του Συμβουλίου θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο έχει πολύ νόημα για τους σημερινούς καταναλωτές. Κάποια, κάποιες παρεξηγήσεις, ε, η ουσία της πρότασης είναι το στο πεδίο εφαρμογής, πακέτα ε, έναντι συνδυασμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ε, δεν είναι, δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει διάκριση στην πρόταση μεταξύ των δύο και θέλουμε ειδικότερα να επιμείνουμε στο γεγονό ότι υπάρχει μια πολύ σαφή ε, υποχρέωση στην πρόταση για τον πάροχο τη υπηρεσία να ενημερώνει τον καταναλωτή τι ακριβώ προσφέρει. Είναι ένα πακέτο και τι συνεπάγεται αυτό το πακέτο ή είναι μια συνδυασμένη ταξιδιωτική υπηρεσία και τι συνεπάγεται αυτό. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι έχει προσφέρει έναν τρόπο να δώσει τη δυνατότητα επιλογής για το επίπεδο προστασίας στον καταναλωτή. Και υπάρχει βέβαια και ένα ε, στοιχείο που αφορά την τιμή. Για τα πακέτα προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε το κόστος ε, σε σύγκριση με το κόστος που έχουμε να αντιμετωπίσουν σήμερα οι καταναλωτές ε, αν, αν επιλέξουν τα οργανωμένα πακέτα και νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό να είναι καλά νέα. Το πακέτο πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο επίπεδο προστασίας, 10 ε, ε, ευρώ ανά που είναι πολύ χαμηλότερο από την ασφάλεια ε, που μπορεί να βρει κανείς σε, οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε ιστότοπο οργάνωσης ταξιδίων αν έχουμε στοιχεία που μας λένε σήμερα ότι αν εσύ είσαι ο άτυχος ταξιδιώτης που αγόρασε ένα πακέτο και αντιμετώπισε ε, πρόβλημα, αν είχε κανείς ε, ε, ακυρώσει κάτι, δεν θα επιβαρυνθεί με κόστος πάνω από το 20-25% της αρχικής τιμής. Δηλαδή, έτσι βελτιώνεται κάπως η κατάσταση για αυτόν τον καταναλωτή. Αν όμως ε, είσαι ένας άτικος ταξιδιώτης ε, ενός άλλου είδους πακέτου, θα πρέπει να επιβαρυνθείς με το 80-85% του κόστους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι φορείς που ήδη εφαρμόζουν τα στοιχεία της ε, οδηγίας. Υπάρχει λοιπόν ήδη κάποιο επίπεδο προστασία. Όσον αφορά το επίπεδο εναρμόνιση, όπω φαντάζεστε, ήταν ε, εσκεμμένη επιλογή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ορίσει το επίπεδο προστασία, γιατί πιστεύουμε ότι λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτή τη επιλογή είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί με εσά, ε, με τα κράτη-μέλη, ε, διάταξη προς διάταξη. Υπάρχουν τομείς για τους οποίους πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να πάμε σε πλήρη εναρμόνιση και άλλους τομείς, και άλλοι τομείς για τους οποίους θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ευελιξία. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα βρούμε μια εξισορροπημένη λύση και ως προς αυτό. Επίσης προσπαθούμε να συσχετίσουμε όντως την οδηγία αυτή με τα δικαιώματα των επιβατών και των επιβατών ε, αεροπορικών εταιριών. Αυτή τη στιγμή αφήνουμε την επιλογή ε, στον ε, επιβατή επιβάτη να απευθυνθεί ας πούμε σε περίπτωση προβλήματος είτε στον ε, οργανωτή του ταξιδίου είτε στην αεροπορική εταιρεία όταν θα συζητήσουμε διάταξη προς διάταξη την, κατά, την, ε, την ε, οδηγία νομίζω ότι θα δούμε ότι έχουμε ένα έγγραφο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε καλή δουλειά για να δώσουμε τη δυνατότητα κατάλληλου επίπεδου προστασίας στους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά και ο εισηγητής μας θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ε, ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ε, δεν χρειάζεται να μας πει τι θα κάνει ακριβώς, αλλά θα πάντων δώσω το λόγο για να μας προετοιμάσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας που ήρθαν και μας μίλησαν με τόση σαφήνεια και ειλικρίνεια και τους συναδέλφους για τις διευκρινιστικές ερωτήσεις που γέννησαν και άλλα ερωτήματα αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσήλωσή της. Ένα όμως κατέστη σαφέστατο από όλους τους ομιλητέ που ακούσαμε. Είναι ευρύτατο το πεδίο όσο και περίπλοκο το θέμα που μας απασχολεί, με πάρα πολύ διαφορετικούς ενεχομένους και πολλά ερωτηματικά που πρέπει να απαντήσουμε. Με ενδιαφέρον θα περιμένω τις συγκεκριμένες προτάσεις και τροπολογίες σας και από πλευράς των εμπειρογνωμόνων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και πραγματικά βλέπουμε σε πόσο σύντομο διάστημα εξελίσσονται τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τόσο γρήγορα, τόσο ραγδαία και πρέπει να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα και όλοι οι ενεχόμενοι ε, να συμμετέχουν με τις προτάσεις τους. Και όλα αυτά όσο γίνεται με χαμηλότερη επιβάρηση από γραφειοκρατική σκοπιά. Να σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχω στη διάθεσή μου που έχει τυπωθεί προς το παρόν. Σήμερα ήταν η ακρόαση και προβλέπεται ήδη 21η ενδεκάτου για, ε, ε, για την έκθεση για να τη στείλω στη μετάφραση. Δύο εβδομάδες. Ε, νομίζω είναι πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα με τόσο υλικό. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο και τους συντονιστές να το ξανασυζητήσουν αν υπάρχει δυνατότητα. Είναι πολύ μικρό το διάστημα. Μέση Δεκεμβρίου παρουσίαση της έκθεση στην Επιτροπή μας και την επομένη 18-12 του λέει λίγη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για να γίνει συζήτηση μέσα Ιανουαρίου στην Επιτροπή και η ψηφοφορία στις 11 Δευτέρου στην ΙΜΚΟ. Μα έχουμε λίγο χρόνο για την έκθεση. Πρέπει να την κάνουμε σε δύο εβδομάδες. Δεν υπάρχει ένα περιθώριο. Δεν μπορώ να το καλύψω μέσα σε δύο εβδομάδες άρον-άρον ε, ε, και μετά τρεις μήνες για συζητήσεις και τροπολογίες. Πώς θα γίνει. Ε, επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να εργαστούμε σε βάθος και με προσοχή και με μέθοδο γιατί θα πρέπει να ισχύσει άλλα 25 χρόνια και να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα και να τα ρυθμίζει. Και αποκλείεται να προκάνω μέσα σε δύο εβδομάδες. Σας το λέω. Κατά τα άλλα, χαίρομαι για το θέμα αυτό και για τη συνεργασία και για τη σύνδεση που κάνουμε με τα δικαιώματα των επιβατών γιατί υπάρχουν συνάφειες και αλληλεπικαλύψεις και συνάντηση, βεβαίω το είπαν και πολλοί προλαλήσαντες και χρειάζονται καθαρές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και πάλι όλους τους ε, συμμετέχοντες. Περιμένουμε χαρά τα σχόλιά σας επόμενα και παρακαλώ αυτά που θα, θα μου δώσετε ως προτάσεις να είναι συγκεκριμένα όσο γίνεται. Δεν χρειαζόμαστε πια γνωματεύσεις 150 σελίδες αλλά συγκεκριμένες ε, προτάσεις για τα διάφορα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να ξαναλάβω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ακρόαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και περιμένουμε ότι θα συνεχίσετε να ασχολείστε ενεργά με αυτό το τόσο ενδιαφέρον ε, θέμα. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω Όσοι δεν ε, θέλουν να παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας για το σύστημα e-call, πάρα πολύ ενδιαφέρον σύστημα, να αποχωρήσουν ε, χωρίς να κάνουν φασαρία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε συζητήσεις έξω από την αίθουσα, να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Πρέπει να δώσω και το λόγο στην κυρία Σενάλοβα να μας παρουσιάσει τις δύο εκθέσεις της. Λέω να μας τις παρουσιάσετε και τις δύο μαζί, να τις εξετάσουμε ως πακέτο. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια γραμμή για τις δύο εκθέσεις. Κύριε Σφάμπ, ε, εκπροσωπείτε τον κύριο Φαντεκάμπ σήμερα. Ο κύριος Μάντερς είναι εδώ, η κυρία Ρούλε είναι εδώ και, ο κύρι... και εγώ είμαι εδώ, μόνο ο σκιώδης συγητής του ΕΛΚ Λοιπόν, η κυρία Σενάλοβα ήταν και η συγγήτρια για την αρχική μας ε, έκθεση πρωτοβουλίας, οπότε έχει πείρα. Είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε συνήθως όταν θέλουμε να ε, αποκτήσουμε κάποια εμπειρία για μια μελλοντική νομοθετική πρόταση. Συνεργαζόμαστε βέβαια πολύ στενά και με την ε, Επιτροπή Μεταφορών γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να μείνω για όλη τη συζήτηση. γιατί πρέπει να πάω και στην Επιτροπή Μεταφορών να τους ε, ε, εξηγήσω τι έγινε στον τριμερή διάλογο για τις ε, επιθεωρήσεις φορτηγών στα οδικά δίκτυα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το e-call, είναι ένα θέμα αρμοδιότητας της δικής μας επιτροπής. Θα αναφερθώ και στην απόφαση για, την, για το σύστημα e-call, ε, μια γνωμοδότηση που είναι αρμοδιότητος της Επιτροπής Μεταφορών. Σήμερα το πρωί έγινε η παρουσίαση και σήμερα είμαι εδώ να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου, τη γνωμοδότησή μας. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τον εισηγητή της Επιτροπής ε, ε, Μεταφορών τον κύριο Ντεμπάκερ ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη. Όπως είχε γίνει άλλωστε και με την έκθεση πρωτοβουλίας μας. Εχθές μόλις το Συμβούλιο είχε την πρώτη συζήτησή του για την νομοθετική αυτή πρόταση και χαίρομαι γι' αυτό Καθυστερεί όμως πάρα πολύ το Συμβούλιο, οπότε πρέπει να πιέσουμε περισσότερο ώστε αυτό το πολύ χρήσιμο σύστημα ασφαλείας ε, να μην καθυστερεί κι άλλο. Να σημειώσουμε πρόοδο. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να εξοπλίσει τα οχήματα με εντός οχήματος συστήματα από τον Οκτώβριο του 2015 για το e είναι κάτι το οποίο επιδοκιμάζω γιατί συνάδει με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη εγκρίνει εμείς Οπότε να προτείνω απλώς ε, κάποια βασικά στοιχεία. Θα αναφερθώ σε βασικές πτυχές, ε, στις οποίες πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την πρόταση. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής. Πιστεύω ότι στο πρώτο στάδιο η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να υπάρχει μόνο στις κατηγορίες των οχημάτων ε, όπου υπάρχουν ήδη κάποιοι μηχανισμοί δρομολόγησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενθαρρυνθεί, να προχωρήσει λίγο παραπέρα και να υποβάλει μία πρόταση ώστε να επεκταθεί η διάταξη e-call για να καλύψει και άλλες κατηγορίες οχημάτων όπως είναι οι μοτοσικλέτες, ε, τα πούλμαν, τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Νομίζω ότι το σύστημα e-call πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εν λόγω οχήματος και επειδή τώρα αναθεωρούμε τις διατάξεις για τις ε, τεχνικές ε, ε, επιθεωρήσεις, νομίζω την ευκαιρία να αναφερθούμε στο 112 τον αριθμό που θα χρησιμοποιεί το e-call ώστε να μπορούν ε, οι δύο μηχανισμοί να λειτουργήσουν παράλληλα, νέα. εξασφαλιστεί η συνέχεια του συστήματος και ε, η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων. Το να χρησιμοποιείτε λοιπόν το 112 ως αριθμός ε, κλήσης για το e-call νομίζω ότι είναι βασικό στοιχείο γιατί τα, οι κλήσεις e-call θα θεωρούνται κλήσεις προτεραιότητας που θα πρέπει να απαντηθούν πρώτες. Όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες, θα πρέπει να υπάρχει μια τηλεματική πλατφόρμα η οποία βέβαια θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές και περαιτέρω για μελλοντικού και περαιτέρω μηχανισμού που θα βασίζονται στο e-call. Κάτι τέτοιο όμω δεν πρέπει να καθυστερήσει την εισαγωγή του συστήματο e e-call, γιατί αυτό είναι πραγματικό ένα σύστημα ασφάλεια προτεραιότητα για μα. Και εμεί θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της ε, ναι μεν οι υπηρεσίε πρέπει να έχουν ε, προστιθέμενη ε, αξία, πρέπει όμως και να συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ε, μία ακόμη σημαντική ομάδα διατάξεων που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι βασική διάταξη για τους ε, τελικούς καταναλωτές. Ας μην ξεχνούμε ότι το e-call βασίζεται σε μία τεχνολογία η οποία δεν επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης του οχήματος, τον εντοπισμό του οχήματος και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Για την ασφάλεια δικαίου λοιπόν, την ασφάλεια δικαίου της ε, συγκεκριμένης πρότασης θα ήθελα ορισμένα πράγματα να αλλάξουν και μιλάω για τις κατεξιοδότηση πράξης, άρθρο 8 συγκεκριμένα, που αναφέρεται στις ε, Εξαιρέσει. Αυτές οι εξαιρέσεις ορίζονται πολύ αόριστα κατά την άποψή μου και θα ήθελα οι ορισμοί αυτοί να αποσαφινιστούν ε, να ξέρουμε ποιες εξαιρέσεις συγκεκριμένα προτείνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα τη γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Μεταφορών, Μιλάμε για την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος e-call σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα διαλειτουργικό σύστημα ε, συντονισμένο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που βεβαίως με βρίσκει σύμφωνη απολύτως και όσες τι χώρες δεν το έχουν κάνει ακόμη θα έπρεπε να το κάνουν ε, πριν από την 1η Οκτωβρίου 2015 το αργότερο. Πρέπει λοιπόν να εισαγάγουν ε, αυτές τις, αυτή την υποδομή ε, επιγουσας κλήσης e-call Νομίζω ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εισαγωγή της τεχνολογίας αυτής που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές ε, θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω στην προθεσμία αυτή. Υπάρχει επίσης και το θέμα της διαδικασίας ε, ε, κατά πόσο είναι αποφελές κάτι τέτοιο και για ποιο, ε, να εξηγήσουμε δηλαδή για ποιο λόγο η υπηρεσία αυτή είναι σημαντική και αυτό με βρίσκει σύμφωνη. Θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι είναι δημόσια υπηρεσία το e και ως τέτοια θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους όσους ε, την έχουν δωρεάν. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Στην περίπτωση του κανονισμού η, η πρόθεσή μας είναι να πάμε πολύ γρήγορα, γι' αυτό έχουμε στενές προθεσμίες. 14 Νοεμβρίου για τον κανονισμό και για την απόφαση 7 Νοεμβρίου. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή mm. κιόλας. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, συναδέλφους να το λάβουν αυτό υπόψη και να ολοκληρώσουν τις ε, τροπολογίες τους. Ε, στις 28 Νοεμβρίου, κατά τη δική μας συνεδρίαση, μπορούμε να οργανώσουμε μία μήνυα ακρόαση. Κάποιοι πυρογνώμονες μπορούν να προσκληθούν και να μας εξηγήσουν κάποιες πτυχές που δεν είναι σαφείς ακόμη σε σχέση με τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Είχαμε κάποιες ακροάσεις ε, ε, στο πλαίσιο της δικής μας, ε, της έκθεσης πρωτοβουλίας μας. Αν έχουν όμως οι συνάδελφοι προτάσεις ή ερωτήσεις, ευχαρίστω να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να οργανώσουμε μια μίνι ακρόαση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως Αναμένω εναγωνίως τα σχόλιά σας και μια πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης συγητές και τους συναδέλφους από την Επιτροπή αυτή, αλλά και από άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σενάλοβα για την ε, πολύ καλή σας παρουσίαση και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των τροπολογιών. Κύριε Σφάμπ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι εκτελώ χρέη και όδους ε, εισηγητή από πλευράς ΕΛΚ, διότι είδατε ότι απουσιάζει ο δικός μας εισηγητής, αλλά τον εκπροσωπώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σενάλοβα, πολύ ε, καλή η πρότασή της, μας βοηθάει πάρα πολύ Ακούω για το χρονοδιάγραμμα ότι είναι πολύ σφιχτό. Ξέρετε, τις επόμενες εβδομάδες θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, όλοι οι συγητές και σκιώδες συγητές. Αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Τι να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να αποφύγουμε τα διάφορα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν. Σήμερα εκπροσωπώ το Wim van de σκιώδη συγητή του ΕΛΚ. Ε, Ζητεί συγγνώμη για την απουσία του. Μία ερώτηση μου ανέθεσε να κάνω για το e-call, αν υπάρχει δυνατότητα εντός της προτάσεως αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να ε, ανατρέχουν και στην ιδιωτική πρωτοβουλία για να έχουν πρόσβαση σε αριθμούς ε, τηλεφωνικής κλήσης ε, για έκτακτη ανάγκη και επίγουσα ή μόνο το 112 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή θα είναι η υποδομή. Είναι πρόβλημα αυτό. Μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Σενάλοβα, πώς θα γίνει η αλληλεπίδραση του συστήματος που υπάρχει ήδη και λειτουργεί και έχει την ίδια διασύνδεση με το 112. Πώς το βλέπει αυτό να γίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεχίσει αυτό το σύστημα. Αυτή είναι η μόνη ερώτηση που έχει ο Βιν ε, Φαντεκάμπ και με επιφόρτησε να τη διαβιβάσω στην εισηγήτρια. Σταματώ αμέσω, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη προσοχή που δώσατε στη σύντομη παρέμβασή μου στα αγγλικά. Okay. Um, well, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και θα ζητήσω από, τις, από το γραμματέα να ε, καταγράφει τις ερωτήσεις. Η κυρία Σαναλόβα έπρεπε να πάει σε άλλη επιτροπή, αλλά υπάρχουν και οι υπηρεσίες της Κομισιόν. Η κυρία Σανάλοβα έχει κάνει κάποιες ε, τροπολογίες, έχει υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες. Μάντους, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την ε, σκληρή δουλειά και για τη συνεργασία. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, είναι εφικτό στηριζόμενος σε αξιολόγηση του 2008, έχουν περάσει πέντε χρόνια και, και ε, εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι παλιό. Μήπως αυτές οι, ε, οι μελέτες αντικτύπου να γίνονται κάπως ε, πιο γρήγορα, τέλος πάντων, να, είμαστε, να προχωράμε μαζί με την εποχή. Εδώ έχουμε το κινητό, ένα κινητό, το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε και να ε, λειτουργήσει στο τηλέφωνο, στο αυτοκίνητο. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα, ένα κουμπί, ας πούμε, on-off, γιατί κάποιος, ας πούμε, θέλει να διατηρήσει την, τον ιδιωτικό του χώρο. Και μετά τι γίνεται με το GPS. Ε, γιατί τότε, ξέρω εγώ, με τους Αμερικανούς σου μπορεί να διατηρήσει κανείς τον ιδιωτικό σου χώρο, ας πούμε, την ιδιωτική σου ζωή. Τι, προφανώς θέλουμε να την ε, προστατεύσουμε, αλλά μπορούμε. Ναι, ε, να σας πω, πρέπει να είστε ευχαριστημένος αν οι Αμερικάνοι σας παρακολουθούν, διότι αυτό σημαίνει ότι είστε μεγάλη προσωπικότητα. Η κυρία Ρούλε. Ναι. Θα σας εκπλήξει ότι μπορεί να συμφωνώ εδώ με τον κύριο Μάντερς. Και εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να σώζονται ζωές, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει ε, να πούμε ότι είναι καλύτερο ένα εθελοντικό σύστημα ε, από ένα δεσμευτικό υποχρεωτικό. Το χάσαμε αυτό στην Επιτροπή, τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα οι χρήστες να έχουν αδιακόπτη, να το ανάβουν και να το σβήνουν να υπάρχει η δυνατότητα από τον κατασκευαστή, ε, αν θέλει ο οδηγός να απενεργοποιεί το σύστημα ηλεκτρονικής κλίσης, να μπορεί να το κάνει. Είναι σημαντικό και μόνο έτσι θα συμφωνήσω. Για μένα είναι κόκκινη γραμμή. Επίσης, έχω και προβλήματα με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους, όπως ο κύριος Μάντερς. Η οδηγία ε, θα πρέπει να αναφέρεται όχι μόνο για την προστασία των δεδομένων όχι μόνο σε αιτιολογικές σκέψεις αλλά και στα άρθρα και να τηρείται ανα πάσα στιγμή και να γίνεται σεβαστή. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πρόκειται για επιπλέον υπηρεσίες γιατί συχνά το βλέπουμε και αυτό. Ε, τηλεφωνούν σε συνεργεία αυτοκινήτων τα οποία κρατάνε τα δεδομένα σου. Ε, αυτό δεν είναι έκτακτη κλίση. Θα πρέπει τελικά ε, ο, ο χρήστης να αποφασίζει σε ποιον θα διαβιβάζονται, αν διαβιβάζονται τα στοιχεία του και ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και βασικές ε, αφετηρίες και αρχές και πρέπει να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζω, επόπτης προσωπικών δεδομένων έχει γνωμοδοτήσει. Ε, μήπως να μας το δώσετε και μας αυτό. Γιατί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και όλο αυτό το ζήτημα έχει σημασία τεράστια σε μια τέτοια οδηγία και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. I think, um... Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι κατάλαβα το σύστημα ενεργοποιείται όταν ενεργοποιηθεί ο αερόσακος. Από ό,τι κατάλαβα, Επαναλαμβάνω, το σύστημα αυτόματα ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται ο αερόσακος. Δεν είναι συνεχώς ενεργοποιημένο το σύστημα δηλαδή. Γιατί πολλές φορές μπορεί να είσαι και να έχει λιποθυμίσει όταν ανοίγει ο, ο, ο, αερόσακος. Άρα εγώ θα, θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι θα ανοίξει. Γιατί ούτω ή άλλω και υπάρχει και η περίπτωση απενεργοποίηση του αερόσακου, αλλά στην θέση του, του, του συνεπιβάτη. Ποτέ δεν απενεργοποιείται στη θέση του οδηγού. Τέλο πάντων, νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Ε, ίσως υπάρχουν, μπορεί, πρέπει να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά τέλος πάντων, καταρχάς πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει απόλυτα δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να είναι συμβατό με τον Γαλιλαίο. Το πρόβλημα είναι πότε θα λειτουργήσει το πρόγραμμα Γαλιλαίους και, πότε, και πόσο θα κοστίσει να γίνει συμβατό με τον Γαλιλαίο. Επί του παρόντος έχουμε ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται κυρίως στην πληροφορία, αλλά όσον αφορά την, ε, το γεωγραφικό εντοπισμό της κλίσης θα χρησιμοποιούμε το GPS. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, συμφωνώ με την παρατήρηση που έκανε ο κύριος για την διαλειτουργικότητα, διότι, πιστε... ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν ένα σύστημα όπου οι οδηγοί μπορεί να έρθουν σε επαφή μαζί τους σε περίπτωση κάποιου περιστατικού. Υπάρχει όμως και ένα ευρύτερο θέμα. Αυτές οι προδιαγραφές για την ε, κατασκευή μιας μονάδας πότε θα είναι ε, διαθέσιμες διότι ας πούμε μπορεί κάποιοι καταναλωτές να θέλουν να ενσωματώσουν το σύστημα αυτό στο αυτοκίνητό τους ήδη όπως είπε ο κ. Μάντρες που να χρησιμοποιούν και το κινητό τους δεν λέω αλλά υπήρξε και μία πρόταση ότι η, η, τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική λύση για το e-call το, e-commission το απέκλεισε αυτό, διότι πολλές φορές οι, έχουν οι καταναλωτές τα, ε, οι οδηγοί τα κινητά τους μαζί. Ή άλλοι να αρχίσει να είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμο το σύστημα. Αυτό θέλουμε. Πάντως καλό θα είναι να υπάρχουν προδιαγραφές έτσι ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί αυτό το σύστημα και ε, να το αγοράσουν αυτοί που ενδιαφέρονται. Λοιπόν, η Μπενεντέτ θέλει να ε, κάνει μια παρατήρηση και μετά θα ήθελα να δώσω λόγο στον κύριο Καραμίτσο και στον κύριο Πετσινέλη να κάνουν κάποιο σχόλιο. Πάρα πολύ σύντομα, μια και η Όλγα Σενάλοβα δεν είναι εδώ, αλλά το έχω συζητήσει μαζί της και βρίσκω και τις απόψεις μου στην γνωμοδότησή της, την ευχαριστώ για αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εποφεληθούμε από το e-call για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και γεωγραφικά τις κλήσεις των smartphones. Δεν γίνονται πολλά πράγματα από πλευρά της Κομισιόν. Όμως οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν τηλέφωνα με GPS ε, συμβατά με την με τους τρόπους γεωγραφικής, ε, γεωγραφικού εντοπισμού. Ούτως ή άλλως ε, μπορούν μέσω της κινητής ε, τηλεφωνίας ο γεωγραφικός εντοπισμός της κλήσης να μεταδοθεί στο 112. Άρα με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη διαφύλαξη του ιδιωτικού βίου των καταναλωτών όπως το ζήτησε και η Τραν και η Ήτρε, θα πρέπει η πρόταση αυτή να ε, εξεταστεί σε συνεργασία, αν θέλετε, και με τις άλλες προτάσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Ε, αν όχι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Καραμίτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την πρόταση ιδίας πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ την κυρία Σανάλοβα και τον συνάδελφο από την Επιτροπή Μεταφορών. Υπάρχει το θέμα και του κέντρου διαχείρισης των κλήσεων αυτών. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, μέχρι τον Οκτώβριο 2015 θέλουμε να το κάνουμε λειτουργικό το σύστημα, άρα το θέμα του χρόνου είναι σημαντικό. Είμαστε πεπισμένοι, όπως και ο εισηγητής σας, ότι το σύστημα αυτό έχει πλεονεκτήματα. Πέρυσι είχαμε 500.000 τραυματίες και 20.000 νεκροί και ε, οι, οι, οι, οι νεκροί ε, πεθάναν ε, μετά την, το ατύχημα. Άρα, ε, σε ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 50%, μπορούμε να βελτιώσουμε την, την έκβαση. Διότι αν μπορούμε να εντοπίσουμε το όχημα, τότε μπορούμε να ενημερώσουμε και τις, τα ασθενοφόρα κτλ. Βέβαια, τα, υπάρχοντα συστήματα έχουν πολύ, μικρά, πολύ μικρή δίσδυση στην αγορά και πιστεύουμε ότι αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν στην πρόθεση του συστήματος που είναι τόσο ε, εποφελές για τους καταναλωτές. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτά τα ότι αυτές, αυτά τα συστήματα ε, ε, είναι μονάχα για λίγους. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε για πολλούς. Αυτό το οποίο προτείνει η κυρία Σελανόβα μπορούμε να τα αφήσουμε ως έχει. Δεν νομίζω με τις ε, τροπολογίες δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο. Απλώς αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω είναι η πλατφόρμα τηλεματικής που ανέκυψε και στη ζήτησή σας ε, εδώ και καιρό που θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και τώρα με τρεις ε, με, το, με τους ταχογράφους, το e-call και το, ε, τα ηλεκτρονικά διόδια μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την τηλεματική πλατφόρμα όπου μπορούμε να, να προσθέσουμε και άλλα πράγματα και με τον Γαλιλαίο που ελπίζουμε ότι θα είναι λειτουργικός ε, γρήγορα γιατί του χρόνου θα εκτοξευθούν οι 14 συνοματικοί δορυφόροι, τότε θα έχουμε ένα πλήρε σύστημα. Κάτι άλλο το οποίο ανέκυψε στη συζήτηση είναι η απενεργοποίηση του συστήματος. Δεν είναι να απενεργοποιηθεί το σύστημα. Το σύστημα είναι, γίνεται, ενεργοποιείται από τη στιγμή που κάποιος σένσορας ε, λειτουργήσει. Μπορεί να είναι ο σένσορα του, του αερόσακου, όπω είπατε πρόεδρε, κάτι τέτοιο. Και τότε ενεργοποιείται το σύστημα. Και υπάρχει ένα κουμπί βέβαια επίση, ε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, κάποιο άλλο περιστατικό. Αν αισθάνεσαι ότι θα πάθει καρδιακή προσβολή και δεν έχει γίνει ατύχημα, τότε πατά το κουμπί. Λοιπόν, ενεργοποιείται το σύστημα μόνο σε περίπτωση του σένσορα, είπαμε και θα ήθελα να το δώσω το λόγο στον συνάδελφο, ο οποίος θα ασχοληθεί με τα θέματα έγκρισης, ο κύριος Πετινέλη. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να δώσω, κάποιες, να δώσω απαντήσεις σε κάποιες από τις ερωτήσεις που έθεσε η συγκίτρια και οι άλλοι βουλευτές. Καταρχάς, το πεδίο εφαρμογής. Εμείς ε, προβλέπουμε να εφαρμόσουμε το σύστημα αυτό στα ε, ιδιωτικά αυτοκίνητα, στα M1 και MM και επιλέξαμε αυτούς τους τύπους αυτοκινήτων διότι πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία ε, είναι υποχρεωμένα να έχουν αερόσακο. Δηλαδή η υποχρέωση ύπαρξης αερόσακου όπως σας είπαμε είναι, το, είναι η η ανάγκη, είναι η απέτηση, μάλλον είναι η απέτηση για να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Ε, η, μελέτη αντικτύπου έχει γίνει με βάση τα αυτοκίνητα που είχαν ήδη ε, αερόσακο. Το να εφαρμόσουμε ε, το e-call σε άλλα μηχανήματα, που, σε άλλα οχήματα που δεν έχει αερόσακο, τότε θα ε, είχαμε άλλο κόστος, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Επομένως είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε μόνο το, σύστημα αυτό, το e-call, στα οχήματα που έχουν αερόσακο. Επίσης, εάν ε, θέλουν ε, να προσθέσουν τα αυτοκίνητα οι αυτοκινητομηχανίες και κάποια άλλα ιδιωτικά νούμερα, αυτό μπορούν να το κάνουν όμως σαν συμπλήρωμα στο 112 το 112 θα είναι ε, διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Υπάρχει όμως και ένα άλλο τεχνικό πρόβλημα, διότι οι κλήσεις ε, του 100, ε, προς το 112 αντιμετωπίζονται <laughs> με προτεραιότητα από τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή αν υπάρχει κάποια συμφόρηση και αν τα ιδιωτικά δίκτυα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις κλήσεις, τα κλήσεις προς το 112 θα περάσουν περάσουν γιατί έχουν προτεραιότητα. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι υπηρεσίες προς τους ιδιώτες αφορούν ε, ας πούμε τα, ε, την, οχηματική, την ε, βοήθεια, την οδική βοήθεια κτλ. Όχι όμως στα ασθενοφόρα. Όμως πιστεύουμε ότι το πιο αποτελεσματικό σύστημα είναι το 112, το πιο, ουσιαστικό, το πιο ε, αποτελεσματικό νούμερο είναι το 112, άρα προς αυτό θα πρέπει να γίνεται η κλίση. Επίσης θα πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα ε, ε, από μόνος του ο οδηγός να απευθύνεται και σε άλλα νούμερα. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η προστασία δεδομένων για αυτά τα συστήματα είναι η ίδια προστασία που προσφέρει και το κινητό τηλέφωνο, το κινητό που κουβαλάμε μαζί μας όλη την ημέρα. Δεν πρόκειται δηλαδή να εκπέμπει αυτό το μηχάνημα τέλος πάντων, το σύστημα κάτι διαφορετικό από ότι είναι κινητό. Τώρα, για το άρθρο 8 και για το e δεν μπορούμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, διότι δεν ξέρουμε τι θα παρουσιαστεί στο μέλλον, αλλά η πρόθεση της Κομισιόν είναι προφανώς να χρησιμοποιούμε το άρθρο αυτό με ένα πολύ ε, περιορισμένο τρόπο μονάχα σε, ε, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο. Παραδείγματος χάρη για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται μόνο στα αεροδρόμια. Εάν μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία ε, κυκλοφορούν μόνο στα, ε, στο, στα αεροδρόμια, τότε δεν χρειάζεται να ε, εξοπλίσουμε το αυτοκίνητο με ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά τέλος πάντων θα υπάρξουν εξαιρέσεις δηλαδή, όμως αυτές οι εξαιρέσεις θα είναι πολύ περιορισμένες. Τώρα για τα σχόλια του Σιώδου Συγητή για τις κλήσεις ε, προς ε, ιδιωτικά συστήματα απήντησα όσον αφορά την ε, ενημέρωση των, της μελέτης αντικτύπου και, την, και τις νέες τεχνολογίες να σας πω ότι για το σύστημα αυτό τα σχόλια ε, ισχύει, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής ισχύουν. Διότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα, για τις ίδιες... Ε, από το 2008 και μετά δεν έχει αλλάξει πολύ η τεχνολογία, διότι μιλάμε για δεδομένα τα οποία μεταδίδονται και με το, με με το κινητό τηλέφωνο. Όπως επίσης τώρα είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ε, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να διότι θα πρέπει όλα τα συστήματα ασφάλειας, το ABS, οι ζώνες ασφάλειας, οι αερόσικοι, δεν μπορούν να ε, απενεργοποιηθούν. Άρα δεν πρέπει να δίνεται δυνατότητα απενεργοποίησης του συστήματος. Έστω και αν υπάρχει θέμα προστασίας ε, των δεδομένων. Τώρα, για το σύστημα Γαλιλαίου, για το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Οι τέσσερις δορυφόροι του Γαλιλαίου που ήδη είναι στο διάστημα εκπέμπουν ένα μήνυμα ήδη. Άρα υπάρχει η αρχή και οι, τα μηχανήματα ή κόλ θα έχουν ένα τσίπ το οποίο θα τους επιτρέπει να ε, λαμβάνουν τα μηνύματα από τον Γαλιλαίο. Το συμπληρωματικό κόστος θα είναι ελάχιστο. Επομένως, μπορούμε να εξοπλίσουμε το σύστημα έτσι ώστε να δέχεται τα μηνύματα Γαλιλαίου, έτσι ώστε όταν το σύστημα γίνει απόλυτα λειτουργικό, να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και για τα e-call. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τα handset ε, και στα, στο αυτοκίνητα αντί για το e-call, αυτή η πιθανότητα είχε εξεταστεί αρχικά, αλλά δεν έγινε αποδεκτή, διότι δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορούσαμε ε, να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα έχουν ένα κινητό μαζί τους, ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα, θα έβαζαν ε, το, το τηλέφωνο, το κινητό τους στην κατάλληλη θέση για να μπορούν να το κάνουν, να κάνουν το e-call και από την άλλη πλευρά τα τρέχοντα τηλέφωνα τα εμπορικά τηλέφωνα δεν έχουν αυτή την αντοχή σε περίπτωση ατυχήματος έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν e-call από μόνα τους. Εδώ νομίζω ότι απήντησα στις βασικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για ε, τις εξαντλητικές ε, απαντήσεις σας. Καλύφθηκαν τα περισσότερα από τα σημεία. Η κυρία Σενάλοβα είπαμε είναι στην Επιτροπή Μεταφορών που έχει και πολλή δουλειά εκεί. Ε, και θέλω να την ευχαριστήσω απουσία τη, Μας έχει δώσει το χρονοδιάγραμμα ήδη για την πρόταση αυτή. Λοιπόν, θα ήθελα να τελειώσει εδώ η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, όπως και εργασίε τη Επιτροπής μας, οι δημόσιε, αν μη τι άλλο. Πάμε αμέσω σε συντονιστέ. Ε, βλέπω ότι είναι παρόντες οι συντονιστέ, Να σας πω ε, την επόμενη συνεδρία που θα είναι 27 Νοεμβρίου, πρωί και απόγευμα, ημέρα Τετάρτη το απόγευμα θα γίνει ακρόαση και πάλι για την πρόταση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δικαιώματα των χρυσών και θα έχουμε την 5η 28 Οκτωβρίου δύο μισές ημέρες πλήρης, 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Ε, να σας ξαναδώ εκεί. Ευχαριστώ για όλους όσους μας παρακολουθούσατε από το διαδίκτυο. Ε, λήξη της συνεδρίασης. Παρακαλώ αποχωρήστε όσο γίνεται πιο σύντομα.